Καλημέρα σας όλοι. Είναι Δευτέρα απόγευμα και πολλοί εκπρόσωποι της, της Επιτροπής μας δεν μπόρεσαν λόγω των αεροπλάνων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αερομεταφορές ε, και δεν μπόρεσαν να φτάσουν, γι' αυτό και είμαστε τόσοι λίγοι. Θα, ε, θα υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη. Και σας ενημερώνω ότι η ψηφοφορία της ε, κατά πρωτοβουλία ε, εκθέσεώς μας για την μείωση της στόχες και δημιουργία θέσεων απασχόλησης αναπτυρώσόμενες χώρες ε, ε, μέθοδος δράσης της κυρίας Θεοχάρους δεν θα ψηφιστεί σήμερα αλλά στις 2 Ιουνίου έχουμε, προτείνει, έχουμε όμως προσθέσει ένα θέμα και η Επιτροπή μας θα γνωμοδοτήσει σχετικά με την έκθεση της νομικής ε, υπηρεσίας για την επιτροπολογία και στην άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όπου έχει καθορίσει συγητή η νομική επιτροπή. Ας προσθέσουμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη ε, και να το συζητήσουμε πριν από τις ψηφοφορίες. Έχετε ε, ένα επιπλέον θέμα ίσως ή συμφωνείτε με τις αλλαγές της ημερησίας διατάξεως. Αν όχι τότε υιοθετείτε η ημερήσια διάταξη. Έχω να σας κάνω μία ανακοίνωση. Η Επιτροπή μας έχει προβλέψει μία αντιπροσωπεία για την Παλαιστίνη. Υπάρχουν δυσκολίες και θα παρακαλούσα τον συντονιστή καθώς και όσους συμμετέχουν να παραμείνουν στην αίθουσα μετά την συνεδρίαση η κυρία Κρετέ, Στράιφλι, ε, Σάιφελτ και ο κύριος Σρέντερ. Νομίζω ότι ε, δεν ε, έχουμε ανακοινώσεις, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα της, ε, των εμποδίων και της και της, των των ατόμων με ειδικέ ανάγκες στις υποανάπτυξη χώρες και σε αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίοι συνήθως αποκλείονται από την αναπτυξιακή βοήθεια. Για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Μουράλι Μπατμακάν ο οποίος εκπροσωπεύει το κονσόρτσιουμ για τις ε, ειδικέ ανάγκες για την κοινή ε, Άννα η οποία είναι εκτελετιστική διευθύντρια της ε, της Επιτροπής Χάνς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πρώτος ομιλητής έχει το λόγο για 7 λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, ε, κυρία Πρόεδρε. Είμαι ο Μουλίμπα Νάμπεντ, ο οποίος εκπροσωπεύει ε, το κονσόρτσιουμ ε, για τα ε, άτομα με ειδικέ ανάγκες και ο οποίος συνεργάζεται ε, εις ε, τον τομέα αυτό. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που, ξε, που μας προσκάλεσε για να Αυτή τη σύμβαση η οποία συνυπεγράφει από τους 27 και οι, ο φορέας μας, η IDDC, ενδιαφέρεται για αυτά τα οποία περιγράφει το σημείο σας και προσπαθεί αυτές τις ιδέες να τις προωθήσει στις 100 χώρες τις οποίες αναπτύσσουν στριότητα. Όσον αφορά τώρα τις ε, αναπηρίες, τις ηθικές ε, ανάγκες, αυτό δεν είναι θέμα μόνο πόσο τυπικό αριθμητικά αποτιμόμενο είναι, ε, θέμα διαφορετικότητας. Η αναπηρία είναι μια αιτία, είναι μια συνέπεια τη φτώχεια, αλλά και η φτώχεια με τη σειράτε είναι συνέπεια και αιτία της αναπηρίας. Επομένως, τα δικαιώματα των αναπήρων είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Και, εγώ όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας, είναι μια κατάσταση επίγουσας ανάγκης η οποία ε, σοβεί. Και τι γίνεται λοιπόν στον κόσμο, τι γίνεται που έχουμε τόσους όλο τον κόσμο οι οποίοι εξαιρούνται, αποκλείονται, περιθωριοποιούνται από όλες τις διαδικασίες της ανάπτυξης. Γιατί όταν έχουμε το θέμα των στόχων της χιλιετίας, εάν θέλετε να πετύχετε με το 2015 στόχο της χιλιετίας χωρίς να βάλετε και εκεί και τους ανάπηρους είναι αδύνατο να μπορέσετε να ελοπίσετε το στόχο αυτό που έχετε τάξει, το στόχο της χιλιετίας διότι έχουμε ε, τόσους φτωχούς οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και ανάπηροι αγαπητοί βουλευτές διότι ε, μιλάμε για το 1 δέκατο του πληθυσμού ένα δέκατο του συνολικού πληθυσμού έχουν κάποια αναπηρία. Επομένως αυτός ο στόχος της χιλιετίας λάβετε το υπόψη. Ποιος, είναι, ποιος ήταν ο πρώτος στόχος, ο επιμέρους. Ε, κρίζωση της φτώχειας. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν βάλετε μέσα σε αυτό το πλάνο και τους ε, ανάπηρους με αντίστοιχα προγράμματα και αντίστοιχες πολιτικές. Κοιτάξτε, τι γίνεται με την παιδεία. Η παιδεία ε, αφορά το 1 τρίτο των παιδιών τα οποία έχουν πρόβλημα αναπηρίας. Μιλάμε για κάποια έκθεση ε, σε παγκόσμια εμβέλεια έγινε και λέει ότι έχουμε 3% της, ε, του αναλφαβητισμού που αφορά τους ε, αναπήρους. όσον αφορά τις γυναίκες έχουμε 1% που είναι ανάπηροι και δεν έχουν αναλφαβητισμό. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να τα κάνουμε όλα αυτά για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για τους στόχους μας, να αγκαλιάσουμε και τους αναπήρους. Υπάρχει επομένω αυτή η σύμβαση, αυτή η συμφωνία του ΟΗΕ που αφορά και τους αναπήρους σε σχέση με την ανάπτυξη. Αλλά τώρα θέλω να σταθώ ιδίω στη διάταξη άρθρο υπαριθμών 4 και ιδιαίτερα την παράγραφο υπαριθμών 3 που μιλά για διαβούλευση και συμμετοχή ε, των ε, αναπήρων εις όλα τα προγράμματα, τα αναπτυξιακά και τις σχετικές πολιτικές. Επίσης έχουμε και το άρθρο 11, το οποίο αναφέρεται στην ανθρωπιστική βοήθεια και σε κάποιες καταστάσεις επιγούσης ανάγκης, οπότε και θα πρέπει και εδώ να ληφθούν υπόψη τα θέματα των ε, αναπήρων. Επίσης έχουμε το 32. και το 32 μιλά για κάποιο είδους συνεργασία δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε αντισιακή συνεργασία εάν δεν καλυφθούν από αυτό το όραμα και οι ε, ανάπηροι. Επομένως με μεγάλη μας χαρά και με ευγνωμοσύνη ε, συμμετέχουμε στη δική σας πορεία μια που εσείς είστε ο μεγαλύτερος δωρητής, δανειστής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει μένως να γίνει διαβούλευση θα πρέπει να υπάρξει mainstream η ένταξη στις πολιτικές, δηλαδή τις πολιτικές για τους ανάπηρους. Θα πρέπει να έχουμε αντίστοιχες καθεντήριες και θα πρέπει να έχουμε την δυτή προσέγγιση ούτως ώστε να καλυφθεί το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, να δούμε τι θα γίνει με τους αναπήρους, πώς θα μπορέσουμε να τους βάλουμε μέσα στο τρένο της ανάπτυξης. Ε, άλλωστε υπάρχει τον Σεπτέμβριο αυτή η συνάντηση κορυφής και θα πρέπει επομένως ε, σε αυτή την διάσκεψη του ΟΗΕ να συζητηθεί ε, το πώς θα προχωρήσουμε προς τους στόχους της χιλιετίας καλύπτοντας, αγκαλιάζοντας και τους αναπήρους. Επομένως, θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τους στόχους της χιλιετίας. Και θα πρέπει να υπάρξει διάλογος με όλες τις χώρες ούτως ώστε να ενθαρρύνουμε την προσυπογραφή και κύρωση της σχετικής σύμβασης του ΟΗΕ αλλά και το προαιρετικό επισυναπτώμενο πρωτόκολλο. Σας ευχαριστώ γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να σας πω τις θέσεις μας και επαναλαμβάνω δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ε, αναπήρους. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα Ας δώσουμε το λόγο στην κυρία Άννα Πελάδ. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Μέλη της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου, επιτρέψατε μου πρώτα-πρώτα να σας ευχαριστήσω ε, εκ μέρους της, του, φορέα, του Ισπανικού Φορέα των Τυφλών, της ΩΝΘΕ για τα θέματα της διεθνούς συνεργασίας και θα πρέπει επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Γερέρο διότι εκείνος ε, πρότεινε ε, αυτήν την ε, πρωτοβουλία όπως έχει γίνει άλλωστε και στο παρελθόν όπως γνωρίζετε αυτή η Εθνική Οργάνωση Τυφλών για την Ισπανία η ΟΝΘΕ είναι ο φορέας που συσπηρώνει όλους τους τυφλούς τώρα τους έχοντες προβλήματα οράσεως στην Ισπανία. Ιδρύθηκε ο φορέα το 1938, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και έχουμε αυτή τη στιγμή 70.000 μέλη. Μέλη οι οποίοι απολάβουν όλων των εξυπηρετήσεων και, και, και, και υπηρεσιών. Ε, βασική μας αποστολή είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε όσους έχουν προβλήματα όρασης να τους εντάξουμε σε όλα τα επίπεδα, σε παιδεία, ε, σε επανένταξη, σε νέες τεχνολογίες, στην κοινωνία της πληροφορίας, σε κουλτούρα, σε πολιτισμό, σε σπόρ, σε αθλητισμό, ε, φτιάξαμε ε, το Ίδρυμα Όνθε. Αυτό το κάναμε για να μπορέσουμε να έχουμε αλληλεγγύη με άλλους ε, αναπήρους, πέραν των ε, οπτικών προβλημάτων. Μιλούμε για 4 εκατομμύρια Ισπανών και, τα βασικά σημεία που μας απασχολούν είναι η επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση και να υπάρχει προσβασιμότητα σε όλα αυτά για όλους τους αναπήρους. Το 98 ε, συνεχίσαμε αυτή μας την αποστολή, αυτή μας την πορεία. Και έτσι ε, ιδρύθηκε το όνθι για την Λατινική Αμερική, ούτω ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε εκεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των τυφλών και όσων έχουν προβλήματα όρασης και στην Ήπειρο εκείνη. Επόμενος, ε, δουλεύουμε σε 19 σπανόφορε χώρες ή, ή τη. Νοτιού Αμερικής, Λατινικής Αμερικής. Τα βασικά θέματα τα οποία μας απασχολούν στη Λατινική Αμερική, <coughs> που γίνεται μέσω της παρουσίας μας αυτές τις 19 χώρες, είναι ε, οι εξή ε, άξονες. Πρώτα-πρώτα, ε, το πώς θα υπάρχει παιδεία που θα καλύπτει όλους ούτως ώστε να καλύπτει όλα τα παιδιά τα τυφλά της Λατινικής Αμερικής και αυτό να το ολοκληρώσουμε σε όλο το 2015. Επίσης, επαγγελματική κατάρτιση, να μπορούν να βρουν δουλειά, να μπορούν να ζουν μια ζωή αξιοπρεπή και, τε, τελευταίο, το να έχουμε την δημιουργία θέσεων εργασίας που να αφορούν τους τυφλούς στην Νότια Αμερική. Τρεις είναι οι βασικές αρχές που μας καθοδηγούν σε όλα αυτά. Πρώτα-πρώτα αυτοκαθορισμό των τυφλών. Α, ε, οπότε ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει οι ίδιοι οι τυφλοί να μπορούν να διαλέξουν, να καθορίσουν το, το, το δρόμο που θα ακολουθήσουν στη ζωή τους και τη διαμορφώσουν ανάλογα. Δεύτερον, έχουμε την ευθύνη του, του, δημοσίου όσον αφορά τις ε, τοπικές αρχές και εθνικές αρχές. Να μην υπάρχουν δεσμενείς διακρίσεις λόγω της αναπηρίας. Κατά τρίτο λόγο, έχουμε κάποια προγράμματα τα οποία να έχουν βιώσιμο χαρακτήρα, να μην εξασφανίζονται μετά τις ε, αρχικές φάσεις. Με αυτή επομένω η παιδεία που θα θέλουμε να τους καλύψει όλους, να σας πω πως, έχει πρώτα πρώτα είπαμε ότι θέλουμε να δούμε πώς γίνεται τόσο ώστε όλοι οι τυφλοί ακόμα και στην, ε, στην, στην, στην Ήπεδρο να μπορούν να πάνε στο γυμνάσιο, να έχουν το, το υλικό που χρειάζονται, την ύλη τους και επίσης για την ε, κατάρτιση κάνουμε ό,τι μπορούμε, προσπαθούμε να του δώσουμε κατεύθυνση, να τους δώσουμε επαγγελματικό προσανατολισμό, ώστε εκείνοι από τους ενηλίκους που δεν είχαν σωστή παιδεία ως νεό και ολοκληρωμένοι να μπορούν να τη συμπληρώσουν όταν ε, ε, ε, βρουν κάποια δουλειά. Οπότε, για την απασχόληση δεν ε, σκοπεύουμε μόνο στο, στην κατάρτιση και στην έβρεση της εργασίας. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε και την αυτοαπασχόληση, κάποιου είδους μικρές προσωπικές ε, επιχειρήσεις, ατομικές και επίσης για το πώς είναι δυνατόν οι θέσεις εργασίας να προσαρμοστούν στα των τυφλών. Και όπου χρειάζεται να υπάρχει και αντίστοιχη επιμελητία και υποστήριξη. Ε, επομένως, ε, επί τη βάση αυτού του ΦΟΑΛ, αυτού του Ιδρύματος. Έχουμε ε, διάφορες ε, επιμέρους υπηρεσίες που μας βοηθούν και επίσης θα πρέπει να κλείσω λέγοντάς σας για το τι λέει για τους αναπήρους ΙΕ. Έχουμε το άρθρο 32 της σχετική σύμβαση του ΙΕ και εκεί λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει διεθνής συνεργασία. Θα πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη, θα πρέπει να υπάρχει απασχόληση, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες πολιτικές. Αυτές που αναπτύσσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τέλει θα πρέπει ως σύσταση ε, προς, τις, ε, προς τα ευρωπαϊκά δημιουργία να σας πω ότι πρώτα πρώτα να αναλυφθεί υπόψη το άρθρο 32 αυτής της ε, σύμβασης όσον αφορά τους αναπήρους. Λέει εκεί ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ανάγκες τους. Τι σημαίνει ληφθούν υπόψη, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εγκάρσια διπλή, διτή προσέγγιση και θα πρέπει επομένω να έχουμε πολιτικές αλλά και προγράμματα τα οποία να έχουν στοχεύσει εις τους αναπήρους. Δεύτερον, πάρα πολύ βασικό θα πρέπει ε, αντί για το φιλανθρωπικό ιατρικό μοντέλο ε, όσον αφορά τους αναπήρους θα πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση που να έχει επίκεντρο τα θεμελιώδη δικαιώματα όλα των ε, αναπήρων, ό,τι ακριβώς ε, ορίζει αυτή η σύμβαση του ΟΗΕ. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του, του, του, των απόψεών μας, να ληφθούν υπόψη ε, οι διαφορετικότητες με, εν μέσω των αναπήρων. Δεν είναι όλοι οι ούτε έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες, ούτε καν έχουν την ίδια αναπηρία. Φυσικά και πρέπει να ληφθούν υπόψη πιο βαριές αναπηρίες, αλλά προσοχή να, νεκριζωθούν οι αιτίε των δυσμενών διακρίσεων. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε ένταξη σε όλες τι πολιτικές, mainstreaming ε, της ισότητας των φύλων. Γιατί και εδώ έχουμε αιτίε δυσμενών διακρίσεων. Να ληφθεί υπόψη. Πέμπτον, να υπάρχει προσβασιμότητα για όλο τον κόσμο. Αυτό να εξασφαλιστεί. Γι' αυτό αφορά ε, ε, ακόμα και τα ίδια τα κτίρια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Εδώ πέρα χρειάζεται να υπάρξει πραγματική και σοβαρή δέσμευση. Έκτον, θα πρέπει να υπάρξουν, να διατεθούν, να δεσμευτούν, να εκταμιευτούν τα χρήματα τα οποία χρειάζονται. Ιδάλω δεν κάνουμε τίποτα. Και έβδομον, θα πρέπει να γίνει σεβαστό ε, το ότι ε, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για τους αναπήρους εάν δεν συμμετέχουν και εκείνοι. Άρα όταν χαράσσονται τέτοιες πολιτικές θα πρέπει να βάλουν υπόψη αυτή η αρχή. Δεν κατακλείδει. Εάν έχουμε ένα κράτος το οποίο ακόμα δεν έχει προσχωρήσει σε αυτή την ε, σύμβαση και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όσο και να το έχουν κάνει αυτό, όσο και αν έχουν ε, κυρώσει αυτή τη σύμβαση, ε, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή και ένα κράτος δεν συμμετέχει δεν θα πρέπει να υλοποιείται το άρθρο 32 και το πνεύμα και οι βασικές αρχές της σύμβασης να μην εφαρμόζονται. Θα πρέπει όμως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ακολουθούν με βλάβια αυτά τα οποία λέει η σύμβαση του ΟΗΕ για τους αναμύρους. Έτσι θα έχουμε έναν κόσμο πιο δίκαιο. Έτσι θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους Ευρωπαίους. Καλύψουν όλους σαν και εμένα και τους ε, συνάδελφους εδώ που μας πήρε. Ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Μπουατάν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της Επιτροπής Αναπτύξεως, Είμαι, ευκαιρία, ευτυχής από την ευκαιρία που μου δίνεται για να απαντήσω στα σχόλια που έγιναν από τις δύο οργανώσεις που πήραν το λόγο και να αναφερθώ στο θέμα των σωματικών αναπηριών στο θέμα της ανάπτυξης. Υπάρχει μία συνθήκη από το Μάιο του 2008 η οποία όμως έχει συναυτεί εν ονόμα της Ευρωπαϊκής Ενώσης μόνο τον Νοέμβριο του 2009 και ακόμη δεν έχουν κατατεθεί ε, τα ε, κυρωτικά έγγραφα ε, βάσει των οποίων θα γίνει η συνθήκη αυτή υποχρεωτική και θα χρειαστεί και ορισμένες προσαρμογές εσωτερικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να μπορέσει να υπάρξει η απόφαση. Εδώ έχουμε ένα ε, σαφές πλαίσιο το οποίο ε, ζητά από όλους τους συμμετέχοντες να καλύψουν τα πάντα οι ε, ε, ε, ε, οι δυνατότητες αυτές συνεργασίες και να προωθηθούν τα, τα δικαιώματα των ατόμων που έχουν σωματικές ανεπάρκειες και αναπηρίες και αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβει και το mainstreaming για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις δράσεις. Έχουμε διάφορες δράσεις από το 2000 ως το 2009 πολλά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν έχοντας σαν βασικό στόχο να βοηθήσουν τις ομάδες των ατόμων με ειδικέ ανάγκες σε διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ε, δυνατότητα ε, αναπτύξεως των προγραμμάτων για άτομα με ειδικέ ανάγκες για να προαχθεί και το νομικό πλαίσιο, αυτό ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ε, διευκολύνουμε την κοινωνική ένταξη σε διάφορες τομείς όπως η παιδεία και η υγεία. Μέχρι στιγμής καλύπτονται οι ανάγκες από τις θεματικές Γραμμέ γραμμές του προϋπολογισμού την ΕΕΣΑΤΕΡ ε ε δηλαδή Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα του ανθρώπου και χρηματοδοτούνται κατά γεωγραφικές ε, ενέργειες αναχώρα και πρέπει να εντάξουμε το δίκαιο των ατόμων με ειδικέ ανάγκες σε όλα τα προγράμματα συνεργασίας πράγμα το οποίο πολλές φορές αποδεικνύεται αρκετά δύσκολο. Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ και στα μέτρα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όχι μόνο για να ε, μειώσει ε, τους περιορισμούς στα άτομα αλλά να μειώσει και την εμφάνιση των ειδικών αναγκών με προγράμματα εμβολιασμού, με καταπολέμηση του AIDS για να μειωθεί το ποσοστό και το σοβαρός χαρακτήρας των σωματικών αδυναμιών που διαπιστώνουμε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο mainstreaming και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της ε, αναπτυξιακής συνεργασίας. Κατά την διαδικασία η οποία είναι η κοινή μας βίβλα, βίβλος δεν αναφέρεται τόσο η σωματική ανικανότητα σαν μία διάσταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αναφέρονται τα δικαιώματα του ανθρώπου αλλά όχι αυτό το θέμα οπότε δεν συμμετέχει ε, το θέμα αυτό στην ανάπτυξη πολιτικών μας όπως άλλωστε αυτό συμβαίνει και ε, για αυτούς οι οποίοι συνεργάζονται για την ανάπτυξη. Επίσης ε, όσο περισσότερο από μακρινόμαστε από την ε, δημοσιονομική ε, ενίσχυση τόσο πιο δύσκολο γίνεται να υπάρξει συγκεκριμένος διάλογος. Γι' αυτό και με τις άλλες χώρες πρέπει να προωθήσουμε την κατανόηση του όρου με τις χώρες αυτές, δηλαδή όταν υπάρχει ένας μειοδοτικός διαγωνισμός που προκυρήσεται π.χ. για άτομα ε, ε, ε, για κτίρια που θα χρησιμοποιήσουν και τα άτομα αυτά πρέπει να προσαρμόσουν οι χώρες αυτές τους κανόνες τους και όχι μόνο αυτούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης υπάρχει ακόμη μία προσπάθεια Ίσως γνωρίζετε ότι στο στατιστικό σύστημα δεν υπάρχει κωδικός για να εντοπίσουμε τις δράσεις που ωφελούν του, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και δεν εμφανίζεται σαφώς αυτό το οποίο γίνεται υπέρ των ατόμων αυτών. Ε, είναι ένα τομέας τον, στον οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε ιδίως στα πλαίσια αυτής της νέας συνθήκης του ΟΗΕ ε, οπότε θα ενταθούν οι προσπάθειες και θα γίνουν πιο κατανοητές. Τελειώνω με ορισμένα συγκεκριμένα θέματα και στα οποία ίσως θέλει να συμμετάσχει και το Κοινοβούλιο. Ξεκίνησε μία μελέτη για τις σωματικές ανεπάρκειες και την προώθηση ε, της ανάπτυξης ε, για να ενταχθούμε στα πλαίσια του προγράμματος του ΟΗΕ. Θα τελειώσει η κατάρτιση του φακέλου στα μέσα του 2010 για να μπορούμε καλύτερα να προσανατολίσουμε τους ανθρώπινους πόρους μας προς αυτό το θέμα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ενημερώσει την εσωτερική guidance note του 2004 επί του θέματος και θα πρέπει να αναθεωρηθεί στα πλαίσια της νέας συνθήκης. Τρίτον, έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργία ενός δικτύου και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης και στις 80 χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε έχουμε εντοπίσει ένα άτομο το οποίο θα είναι ο σύνδεσμος και θα θέλαμε αυτό να καλύψει όλες τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Χάρη στη στενή συνεργασία που έχουμε με το Consortium IDDC που μίλησε προηγουμένως. Βασιζόμαστε σε αυτούς για να προχωρήσουμε και είμαστε στη διάθεσή σας για να ακούσουμε το Συμβούλιο και ε, το Κοινοβούλιο και ε, να καταρτήσουμε τη δράση μας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχουν τώρα οι ομιλητές. Ο κύριος Γκερέρος Σαλόμ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τους ε, δύο εισηγητές που μας ε, παρουσίασαν ε, την δική τους την άποψη του θέματος. Αυτό ισχύει τόσο για την εκπρόσωπο των απείρων όσο και για όλους τους υπολείπους. Για την εκπρόσωπο της ΟΝΣΕ. Η ΟΝΣΕ, η οργάνωση αυτή είναι ένα παράδειγμα το οποίο μπορούν να το κατανοήσουν ε, μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν πάει στην Ισπανία και έχουν δει τι ακριβώς κάνει αυτός ο Ισπανικός ε, φορέας για τους ε, τυφλούς. Ο φορέας αυτός έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για την εκπαίδευση των τυφλών. Κατά το παρελθόν λοιπόν Η οργάνωση αυτή διαδραμάστησε ε, καθοριστικό ρόλο κατά την ε, κοινωνική ενσωμάτωση. Ε, μπόρεσε να βοηθήσει ανθρώπους αυτούς να τύχουν κοινωνικής αποδοχής, να βρουν θέσεις εργασίας. Οι περισσότεροι τυφλοί στην Ισπανία ζουν από δραστηριότητες τις οποίες τους προσφέρει η οργάνωση αυτή, ο φορέας αυτός, ο ΟΝΣΕ. Αυτός ο φορέας πρέπει να πω ότι έκανε τους τυφλούς ορατούς στην Ισπανία. Ο φορέας αυτός έχει μακρά ιστορία ε, στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Έχει αφήσει τα ίχνη του ε, στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στην ίδρυση των διαρθρωτικών ταμείων, στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω επίσης όπως ακριβώς το είπε και η εκπρόσωπος της ΟΝΣΕ, ότι η ΩΝΣΕ δεν παίρνει μόνο μέσα από την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά και η ίδια είναι φορέας χρηματοδότησης και ως εκ τούτου αποτελεί και συνεργάτη της δικής μας Επιτροπής. Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι είναι ε, σάρξ εκ της σαρκός μας. Η ΩΝΣΕ συνεργάζεται με εμάς και συνεργαζόμαστε από κοινού για τη μεταφορά αναπτυξιακής βοήθειας κυρίως στη Λατινική Αμερική. Ε, τώρα λοιπόν για να αναφερθώ λιγάκι ε, στην ΟΝΣΕ και σε αυτά που είπε ο πρώτος μιλητής. Ε, θα πω αυτά που έχουμε πει επανειλημμένα στο Κοινοβούλιο. Η φτώχεια είναι ένα χαρακτηριστικό των τυφλών. Οι τυφλοί είναι διπλά φτωχοί. Και γι' αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής, η παιδεία αυτών των ανθρώπων. Ε, όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν στο να μειωθεί η, ε, η κατάσταση, να βελτιωθεί η κατάσταση των τυφλών, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πρέπει κατά κάποιον τρόπο ε, να γίνουν αυτόνομοι, κοινωνικά αυτόνομοι. Για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ στηρίζω ανεπιφύλακτα το άρθρο 32 της ε, Σύμβασης όπου αναφέρεται ότι όλες οι πολιτικές της ε, αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να έχουν οριζόντια προσέγγιση που καλύπτει και αφορά και στην, στους τυφλούς. Θα ήθελα τώρα να πω κάτι που το ανέφερε προηγουμένως η Κομισιόν. Εγώ Έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτά που στο μέλλον δεν ήταν προφανή θα πρέπει να καταστούν προφανή στο μέλλον. Εφόσον λοιπόν το θέμα είναι να ελέγξουμε τις δύο συμβάσεις που έχουμε υπογράψει, νομίζω θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία για να πούμε ξεκάθαρα κάτι το οποίο δεν ελέγχθη με απόλυτη σαφήνεια το 2005. Οφείλουμε λοιπόν να κάνουμε πρόοδο στην ε, παρακολούθηση των μέτρων, ε, κυρίως όσον αφορά τη συνεργασία ε, σε θέματα αναπτυξιακής βοήθειας. Οφείλουμε να μεριμνήσουμε έτσι ώστε οι οργανώσεις να μπορούν να συμμετέχουν ε, στις μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δικές μας οι αντιπροσωπείες στο εξωτερικό ε, πρέπει να ευαισθητοποιηθούν για να ενεργοποιηθούν και αυτές. Και τέλος θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση στον κύριο Μπάν Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. να μας πείτε τι ακριβώς πιστεύετε για το άρθρο 32. Το άρθρο 32 της ε, Συνθήκης των ΗΠΑ πώς ακριβώς μπορεί να εφαρμοστεί, ε, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε ανθρώπους με αναπηρία και μια, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ή ε, να αντιμετωπιστούν οι τυφλοί στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων. Ο κύριος Γκέρνς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω αυτούς που παρουσίασαν τα θέματα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας υπέδειξε τι δράσεις αναλαμβάνει παρόλο που δεν υπάρχει ευρωπαϊκή συνένεση για την ανάπτυξη είπατε ότι υπάρχουν 300 προγράμματα που τρέχουν. Ε, Υπάρχουν όμως ερωτήματα στρατηγικά. Υπάρχουν οι κρατικοί παράγοντες, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ιδίως η ε, Handicap International. Υπάρχουν τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών και εδώ σκέφτομαι ιδιαιτέρως ε, αυτά τα οποία ε, ξεκίνησαν μετά από το Βιετνάμ που ασχολούνται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται μετά από τις ε, βόμβες που έπεσαν στο Λάος και στο Βιετνάμ και τελικά κατέληξαν εις ε, τις βάσεις της Ταϊλάνδης χωρίς όμως ε, να εκραγεί το αεροπλάνο διότι τα άτομα αυτά έχουν μείνει ανάπηροι 40 χρόνια μετά από τον πόλεμο του Βιετνάμ και θα ήθελα να ξέρω αν έχουμε ασχοληθεί με την οικονομική ευθύνη της χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών διότι ε, εφαρμόζοντας ε, το πρόγραμμα ότι ο Ριπένον πληρώνει θα έπρεπε ε, τουλάχιστον ένα μέρος της χρηματοδοτήσεως να πληρωθεί από αυτούς οι οποίοι προκάλεσαν το πρόβλημα. Το έχουμε σκεφτεί και η σκέψη αυτή έχει προχωρήσει και δεύτερον, ε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια στρατηγική ε, εναλλακτική λύση, δηλαδή ε, αναφερθήκατε στη δυσκολία, στις επιπτώσεις των πολλαπλών, πολλαπλών δράσεων ε, οικονομικής στήριξης. Δηλαδή, εσείς αναθέτετε τους πόρους στη χώρα η οποία την εντάσσει στη στρατηγική της οποίο δεν είναι κατακριτέο, αλλά το θέμα είναι ποιος ασχολείται με το εάν οι ανάγκες αυτές ικανοποιούνται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ποιος συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα, διότι ενδεχομένως μπορούμε να πούμε ορίστε, όπως ε, στα Ηνωμένα Έθνη εμείς θα καλύψουμε ένα μέρος των εξόδων στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο επίπεδο κρατών μελών πράγμα που θα ήταν μια διαφορετική ε, μορφή δημοσιονομικής στήριξης ε, ε, πλέον από μια διεθνή οργάνωση. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους παρεμμένοντες, στον κύριο Παντμαντάν αν επιτιθυμεί, να απαντήσει στους ευρωβουλευτές και στις ερωτήσεις τους. Μικρόφωνο παρακαλώ. Δυστυχώς δεν έχει μικρόφωνο, είναι κλειστό το μικρόφωνο του μιλητή. Λοιπόν, όσον αφορά στο άρθρο 32, στη διεθνή συνεργασία, εκεί προφανώς υπάρχει περιθώριο διαλόγου με τις συνεργαζόμενες χώρες, έτσι ώστε να μπορούν και να ενθαρρυνθούν οι συνεργαζόμενες χώρες να συμπεριλάβουν τους ε, τυφλούς ε, στις ε, δραστηριότητες τους. Γιατί κατ' ουσίαν οι φραγμοί είναι εκείνοι που εμποδίζουν την πρόοδο, έχουμε φραγμό ενημέρωση και βεβαίως και φυσικούς φραγμούς τα ε, μνημόνια της ε, συνεννόησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και θέματα τυφλών. Εγώ τουλάχιστον αυτό πιστεύω ότι ισχύει για το άρθρο 32 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη συμφωνία που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συνεργαζόμενες χώρες. Κύριε Ελαεύ, επιθυμείτε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά το άρθρο 32 της συνθήκης ε, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτό σημαίνει ευθύς εξ αρχής ε, να λαμβάνει κανείς υπόψη του τα δικαιώματα τα οποία αναφέρονται στη Διεθνή Συμφωνία. Όμως ε, αυτό ε, κατ' ουσίαν σημαίνει τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Το μόνο που είναι διαφορετικό σε αυτή τη συνθήκη σε σχέση με άλλες είναι εκείνο που έχει σχέση με την ε, προσπελασιμότητα. Δηλαδή, εκείνο το οποίο θα πρέπει ε, να το αναθεωρήσουμε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε, παραδείγματο χάρη, όλη αυτή την έννοια ατόμων με αναπηρία. Εξάλλου αυτό αναφέρεται και στο άρθρο υπαριθμών 1. Αν διαβάσετε το άρθρο 1 θα δείτε όλη αυτή η κοινωνική, οικονομική δομή ε, στην οποία έχουμε φτάσει. Ο τρόπος ε, με τον οποίο λειτουργεί ένα άτομο με ε, αναπηρία καλείται το άτομο αυτό να λειτουργήσει μέσα σε ένα πλαίσιο με πάρα πολλούς φραγμούς αυτό είναι το θέμα το οποίο νομίζω θα πρέπει να μας απασχολήσει. Θα πρέπει λιγάκι να δείτε και τα στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ανάπηροι. Πολύ σπάνια γίνεται αναφορά σε αυτό. Όταν όμως γίνεται αναφορά, το μόνο που αναφέρεται είναι τα άτομα με αναπηρία σε κάποια κοινωνία είναι ένα σχέριθμος. Το θέμα όμω δεν είναι να δούμε μόνο του αριθμού, να δούμε ποιοι είναι οι φραγμοί που υφίστανται σε μια χώρα, έτσι ώστε τα άτομα αυτά να έχουν τις ίδιες ακριβώς ευκαιριε που έχουν και οι υπόλοιποι πολίτες. Έτσι λοιπόν το άρθρο 32 αναφέρεται ακριβώς σε αυτό. Αναφέρεται σε μία δέσμευση που πρέπει να αναλάβουν τα κράτη-μέλη για να ε, λάβουν μέτρα έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά ε, σε φάση εκκίνησης. Γιατί υπάρχουν διαφορές ακόμα και ανάμεσα ε, στις ίδιες γεωγραφικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου το άρθρο αυτό το 32 θα πρέπει να την υπόψη και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμφίβολα θα πρέπει να προάγουμε τη διεθνή συνεργασία αλλά θα πρέπει ε, και να έχουμε κατά νου ότι όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορούν ε, να καταφεύγουν ε, σε αυτή τη σύμβαση και το ίδιο να ισχύει και για όλους τους ε, υπολείπους. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για να συνοψίσει ο κύριος Μπουαντά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για να απαντήσω σε τρία θύματα που έθιξαν ε, οι ευρωβουλευτές για την ε, ε, προβολή. Ο κύριος Πίμπαλς είπε ότι θα αναθεωρήσει τη συμφωνία του 2005. Όταν θα γίνει αυτό λοιπόν θα πρέπει να, να, υπόψη τις α, τροποποιημένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρώπη και να μπορέσει το θέμα αυτό των σωματικών ανεπαρκειών να συζητηθεί και να γίνει αποδεκτό με την, από νέο πρίσμα. Το ίδιο ισχύει και σχετικά με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που θα συγκεντρωθούν εις την Νέα Υόρκη και να δούμε αν στα προγράμματα αυτά έχουν ε, μείνει στο περιθώριο τα άτομα με ειδικέ ανάγκες στις υποανάπτυξη χώρες. Άρα ε, θα πρέπει να ξαναπροχωρήσουν στο προσκήνιο τα θέματα αυτά. Ε, βεβαίως το θέμα είναι τι θα γίνει αν υπάρχει ε, μια αναπηρία η οποία οφείλεται σε πόλεμο ή σε μια βιομηχανία κτλ. Και πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει εκεί και κατά πόσον είναι συνεκτικές οι αναπτυξιακές πολιτικές διότι όταν είχαμε δεχθεί την οδηγία για το Σεβέζο για σοβαρές αναπηρίες ή όταν ζητούμε να καταργηθούν οι νάρκες εναντίον των ανθρώπων και άλλα μέσα τα οποία βλάπτουν τον άνθρωπο τότε θα πρέπει να εξετάσουμε και τους τους λόγους αυτών των αναπηριών, ε, ιδίως όταν πλήττουν άτομα. Επίσης πρέπει να εξετάσουμε εάν ε, θα υπάρχει ενίσχυση δημοσιονομική ή άλλη. Θα έλεγα όμως ότι εάν περιλαμβάνουμε ε, εις ε, το, εις ε, στα ταμεία μας τις δράσεις οι οποίες είναι ευρωπαϊκές τότε θα μείνουν πολλοί οργανισμοί οι οποίοι δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ενώ αν αλλάξει η εσωτερική νομοθεσία μιας χώρας σαν το Μαλάου ή την Τανζανία για να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε όλα τα παιδιά παραδείγματος χάρη, τότε θα έχουμε μεγαλύτερη απήχηση και όχι μόνο τη χρηματοδότηση των, προγράμμα, προγραμμάτων τα οποία εμείς χρηματοδοτούμε άμεσα. Θα πρέπει όμως να θεωρήσουμε τότε τους αναπήρους σαν μια ομάδα η οποία είναι ένα βασικό ε, στοιχείο της χώρας με την οποία συνεργαζόμαστε και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε καλύτερα να ανταποκριθούμε στην επίλυση του προβλήματος των αναπηριών στον τομέα αυτό. Ωραία. Τώρα ερχόμαστε στο έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως που είναι η εξωτερική εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως. Το περασμένο μήνα είχε παρουσιαστεί ε, μία πρόταση εις ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την περίοδο 2007-2013 ε, με τακτική νομοθετική διαδικασία με διπλή ε, νομική βάση το άρθρο 2012 συνεργασία με τις τρίτες χώρες και, 2009, 209 ε, συνεργασία στα πλαίσια της Ευρώπης όπου θα αναπτυχθεί η πρόταση και ένα βασικό στοιχείο είναι η ενίσχυση της τράπεζας για να μπορέσει να ανταποκριθεί στους αναπτυξιακούς στόχους της ε, Ευρώπης διότι οι περισσότεροι συνεργάτες μας είναι υπό ανάπτυξη χώρα και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μία γνωμοδότηση ο εισηγητής είναι ο κύριος Μπέρμαν και ζητήσαμε να θεωρηθούμε σαν συνδεδεμένη επιτροπή στην ανάπτυξη αυτού του σοβαρού θέματος για το οποίο θα συζητηθεί την άλλη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Έχουμε ζητήσει και μία έκθεση από τον καθηγητή Γκρίφις Τζόνς για την ανάπτυξη, για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως. Έχετε λάβει όλη αυτή την μελέτη, τις οποίες στο φάκελό σας υπάρχει η περίληψη. Γι' αυτό έχουμε καλέσει τον Ντομινίκ Ντεκράιεν Τούρλ, υπεύθυνο για τις θεσμικές υποθέσεις, και τον Τζόρτζο Κιάριαν Κασόνη, ο οποίος είναι υπεύθυνο για το συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή στην Γενική Διεύθυνση ΕΚΒΑ. Δίνω το λόγο πρώτα στον Κιτής Μπέρμαν, ο οποίος είναι ο εισηγητής μας για περίπου 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από αίτημα της Επιτροπής Ανάπτυξης, η Στέφανη Γκρίφιν Τζόουνς παρουσίασε μία έκθεση, μία αξιολόγηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσον αφορά και σε σχέση με την εξωτερική της εντολή, τις αρμοδιότητες που αφορούν στην Ασία, ε, την Νότια Αμερική. Δεν καλύπτει όμως τις χώρες ΑΚΕ, καθότι οι χώρες αυτές ε, καλύπτονται με άλλη εντολή ε, από την Παγκόσμια Τράπεζα. Στέφεν Γκρίφιθ Τζόνς είναι μια πολύ γνωστή οικονομολόγος. Το τελευταίο της βιβλίο το δημοσίευσε μαζί με τον ε, οικονομολόγο Στίγκλιτς. Ε, απλά για να καταλάβετε ποια είναι, έχει πάρα πολύ καλή φήμη. Τώρα, Εκείνο το οποίο υπογραμμίζει στην έκθεση αυτή είναι ότι οι κρατικές τράπεζες καλούνται να διαδραματίσουν συγκεκριμένο ρόλο στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Πρόκειται για έναν αντικυκλικό ρόλο όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Δηλαδή εκεί ε, φαίνεται και η μεγάλη σημασία των τραπεζών. Μπορούν να είναι αντικυκλικές σε περίοδο κρίσης όπου ε, υπάρχει έλλειψη ρευστότητας ε, ας πούμε όταν για τις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχουν ε, πολύ λιγότερα εμβάσματα και όταν υπάρχει και ε, στενότητα στην πίστη. Έτσι λοιπόν οι τράπεζες αυτές μπορούν να λειτουργήσουν αντικυκλικά με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή να στηρίξουν ε, τις ε, καταραίουσες αγορές και εκείνους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι κρατικές λοιπόν τράπεζες μπορούν και πρέπει να διασφαλίζουν το ρόλο τους στο να προσφέρουν την πρόσβαση. Και όπως ε, και οι ιδιωτικές τράπεζες θα πρέπει να παραμένουν ιδιαίτερα αξιόπιστες. Ε, είναι εκείνες οι οποίες κυρίως προσφέρουν μακροπρόθεσμα δάνεια ε, και δάνεια σε σχέση με την αύξηση της ανάπτυξης. Ας δούμε τώρα συγκεκριμένα το ρόλο τους. Σε περίπτωση δημοσιονομικής κρίσης είναι πολύ σημαντικό για μια αναπτυσσόμενη χώρα να της προσφερθούν δάνεια γιατί αυτό όπως ξέρετε πολύ καλά δεν το πράττουν εύκολα οι ιδιωτικέ τράπεζε. Τα κεφάλαια λοιπόν, λοιπόν έρχονται κυρίως από το δημόσιο γιατί ε, στεγνώνουν τα ιδιωτικά δάνεια. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί φραγμοί ε, όσον αφορά τη χρηματοδότηση στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, και ένας φαύλος κύκλος ξεκινάει με την κρίση και επιδεινώνεται με την κρίση. Όπως σας είπα λοιπόν παρουσιάζεται στενότης και έλλειψη ρευστότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες από το 2006 όπως βλέπετε στη διαφάνεια μέχρι το 2007 υπάρχει αύξηση των αριθμών και από το 7 στο 9 τραγική μείωση αν πάμε σε στοιχεία μιλάμε για ε, ροή ιδιωτικών κεφαλαίων 697 δις το 7 και το 9 μείων. 52 δις δολάρια. Δηλαδή εκροή κεφαλαίων από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δηλαδή τι διαπιστώνουμε, διαπιστώνουμε ακόμα και την αντίστροφη ροή. Και το ίδιο, αν θέλετε, ισχύει και για συγκεκριμένες άλλες περιοχές ε, του κόσμου. Η Αφρική που είναι το σκούρο μπλε στο γράφημα που βλέπετε πίσω μου, η Αφρική δεν επηρεάζεται τόσο πολύ από την χρηματοπιστωτική κρίση. Απλά και μόνο γιατί η Αφρική είναι εκτός των ροών. Οι ροές, οι κεφαλαιακές έχουν ήδη πάυσει προς την Αφρική. Ε, στην Ευρώπη βλέπουμε, αυτό είναι το κόκκινο, από το 8 στο 9 είχαμε ε, τραγική μείωση ε, εισρωής κεφαλαίων ή ε, και στις χώρες της Σοβιετικής Ένωσης και εκεί ριζική και ακραία μείωση κεφαλαίων. Βλέπετε λοιπόν ότι τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα αρνητικά για πολλούς ανθρώπους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, αγρότες και ούτω καθεξής. Αν δούμε τώρα τον ρόλο των πολυμερών τραπεζών, πολλές εξ αυτών όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, αύξησαν γρήγορα τις ε, υποχρεώσεις τους. Και έτσι λοιπόν αντέδρασαν ταχύτατα στην κρίση. Η ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αντέδρασε με μικρότερη ταχύτητα. Με υψηλή δανειοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με υψηλή δανειοδιότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές εκταμιεύσεις το 2008. Χαιρετίζω τον κύριο Ντεκρεονκούρ που μόλις μπήκε. Δεν έχω πει τίποτα νέο για σας. Τα γνωρίζετε όλα αυτά. Ήρθατε όμως όταν άρχισαν να κατακρίνω την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γιατί έλεγα ότι ήταν αντικυκλική και ε, δεν, ε, ε, δεν κινήθηκε γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν το βλέπετε αυτό εάν ε, κοιτάξετε τις, ε, την εικόνα αυτή γιατί εδώ βλέπετε όλες τις τράπεζες, την World Bank, την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Ασίας και κάτω έχετε την Αφρικανική Τράπεζα αλλά βλέπετε ότι όλοι αύξησαν την, τα δάνειά τους μεταξύ 2007 και 2009 ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως αύξησε λιγότερο αλλά αύξησε όμως και ότι δεν συνέβησαν πολλά. Αλλά εάν δείτε την ακριβή εικόνα, η, τα δάνεια αυξήθηκαν πολύ για τις προενταξιακές χώρες, τις ανατολικές χώρες και τη Ρωσία ενώ στη Μεσόγειο η κατάσταση είναι διαφορετική. Η ουσία είναι ότι στις προενταξιακές χώρες συνέβησαν πολλά και στις υποανάπτυξη χώρες ε, μειώθηκαν και στις χώρες και ε, τα δάνεια κατά το 2008. Βλέπετε λοιπόν ότι ε, το 2008 ορισμένες δεσμεύσεις ε, σταμάτησαν τελείως και ο όγκος αναπτύχθηκε πάλι το 2009 αλλά όχι τόσο πολύ. Μπορείτε λοιπόν να πείτε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να κάνει περισσότερα και καλύτερα αυτά που πράττει. Ε, θα, θα μπορούσε να αναλάβει περισσότερο κίνδυνο ιδίως για τις χώρες ε, που αξίζουν όπου ε, δεν είναι μεγάλος ο κίνδυνος θα μπορούσε να βοηθήσει πιο ευέλικτα τις υποανάπτυξη χώρες και να συνεργαστεί καλύτερα με τα ε, τους διεθνείς ε, χρηματοδοτικούς θεσμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρειάζεται περισσότερους πόρους. Ενώ κατά την περίοδο της ε, κρίσεως οι δραστηριότητες είχαν αυξηθεί πάρα πολύ και χρειάστηκαν να αφαιμάξουν το προσωπικό ενώ πιστεύουμε ότι αντιθέτως η τράπεζα θα χρειαζόταν ε, περισσότερο προσωπικό για τις ε, εξωτερικές ε, συνδρομές της η οικονομική ένταξη πρέπει να είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος μας δηλαδή να έχουν ε, οι απλοί πολίτες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, οι γεωργοί ε, οι γυναίκες μια οικονομική στήριξη που θα βοηθούσε με μια διερκή πορεία την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα, τον λόγο για ο κύριο Ντεκρανιακούρ για περίπου 7 λεπτά, λέει η Πρόεδρος. Thank you Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να σας πω με δύο λόγια τα βασικά θέματα εκείνα τα οποία απορρέουν από την ονομαζόμενη έκθεση Καμπτουσίου διότι αυτό θα είναι το θέμα στη μέση διάταξη, το οποίο θα μας απασχολήσει εις τους αμέσως επόμενους μήνες. Και θα ήθελα να σας πω τα πέντε βασικά σημεία τα οποία ε, υπάρχουν στο κείμενο εκείνο. Τα περισσότερα από όλα αυτά, αν όχι όλα, περιλαμβάνονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρώτα-πρώτα. Η αποδέσμευση 2 δις από την εντολή αποθεματικού, τόσο ώστε να χρηματοδοτούν αυτά τα προγράμματα για την ε, αλλαγή του κλίματος. Και από ό,τι φαίνεται αυτό πρώτα να πειρώσει και να συγκεντρώσει τη γενική συνένεση του κόσμου. Δεύτερον και πάρα πολύ σημαντικό, ιδίω όσον αφορά την ΕΤΕ, έχουμε το ότι θέλουμε να κάνουμε streamline των ε, βασικών στόχων όσον αφορά την εντολή για τα διάφορα μέρη του κόσμου, γιατί πρώτα απ' όλα τώρα έχουμε ένα, ένα ψήφι δοτό με διαφορετικού στόχου όσον αφορά την κάθε περιοχή, γιατί κάθε φορά εξαρτάται τι ιστορικά έχει κριθεί ότι πρέπει να γίνει. Τώρα όμω όλα θα τα έχουμε πάνω στην ίδια βάση, επί τη βάση τη υποδομή, σαν κριτήριο, τη αλλαγή του κλίματο, ε, τη ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και τον ΜΜΕ, κάτι κατά τρίτον και πάρα πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο έχει να κάνει με την Επιτροπή σας είναι το ότι σκοπός ε, είναι το να μπορέσουμε να τονίσουμε την πτυχή ανάπτυξη αυτών μας των ε, κινήσεων τρίτων και επίσης πάρα πολύ σημαντικό και στο οποίο θα επανέλθω είναι το ότι θέλουμε να υπάρχει προσαρμογή των μέσων εις τους στόχους και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο πρόκειται αυτά τα οποία είπε ο κ. Βέρμαν να τα προσαρμόσουμε δηλαδή του ανθρώπινου πόρου στον στόχο στη δουλειά, ούτω ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε του ανθρώπινου πόρου για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση ε, τη ε, ΕΤΕ σε αυτά τα κεφάλαια, αυτέ τι υποτροφίε ε, για μία σειρά δράσεων, αλλά επίση και για το, να, για το να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποια συνέργεια μεταξύ μας, ε, ούτως ώστε να μπορέσουμε ενδεχομένω να μοιραστούμε και τα ίδια γραφεία των αντιπροσωπιών μα εκτό ΕΕ. Πέμπτον, η αναβάθμιση τη συνεργασία με την Επιτροπή αλλά και με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Θεωρούμε δε ότι η ΕΤΕ είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι από το αντίστοιχο της Κομισιόν όσον αφορά τη χορήγηση αυτών των ε, πόρων, αυτών των κεφαλαίων από τον κοινωτικό προπολογισμό. Και άρα θα πρέπει να μπορεί να έχει κάποια βοήθεια από του εθνικού προπολογισμού, αλλά και από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσον αφορά δηλαδή κάποια δάνεια που προχωρούν παράλληλα με τι χορηγήσει τη ΕΤΕ. Τώρα, ε, αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε απαιτούν επίσης ε, περισσότερη δουλειά, περισσότερη προσπάθεια όπως και το να έχουμε ένα καινούργιο φορέα για να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες και τους πόρους τη ε, της χρηματοδότηση από Κομισιόν και από ΕΤΕ και ενδεχομένως αυτή η καινούργια υπηρεσία να εξελιχθεί σε μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα Συνεργασίας και Ανάπτυξης έτσι να έχουν περισσότερη προβολή αλλά και περισσότερη αποτελεσματικότητα για όλα αυτά τα μέσα τα οποία αυτή τη στιγμή τώρα είναι διασπαρμένα πολυδιασπασμένα σε διάφορα μέσα Ευρωπαϊκή Ένωση άρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να κινηθεί μια διαδικασία και να αρχίσουμε κάποιες μελέτες ε, επιπτώσεων ε, to, adapt... και μελέτες σκοπιμότητας ε, οπότε και πρέπει επομένω να συντεριάξουμε τα μέσα με του σκοπού. Επομένω, όπω είπαμε, όσο περισσότερο κανεί προχωρεί όσον αφορά την πολιτική τη ανάπτυξη, χρειάζεται περισσότερο ανθρώπινου πόρου, χρειάζεται κεφάλαια και διακυβέρνηση ανάλογη. Είδατε στην έκθεση Καμπτεσίου ένα παράδειγμα το οποίο δείχνει αυτό τον λόγο, την αναλογία μεταξύ των ανθρωπίνων πόρων του προσωπικού. Ε, και είδατε ότι υπάρχει εκεί δυσαναλογία αναλογία που φτάνει μέχρι το 1 προς 40 ανάλογα με, με, με, με, τι συγκρίνεται, ποιο, ποιο ίδρυμα, ε, ποιο, ποιο, ποιο θεσμικό όργανο συγκρίνεται με την ΕΤΕ. Ε, οπότε μιλάμε για επιδοτήσεις, μιλάμε για χορηγήσεις, ανάλογα με τους κανόνες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και ε, κάποια εξωτερικά στοιχεία ή κάποια στοιχεία επίσης χαριστικού χαρακτήρα ανάλογα με το τι θέλει να πετύχει. Οπότε, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, έχουμε αυτή την έκθεση των σοφών ε, για, αυτή την, για αυτό το χωριστό νομικό πρόσωπο στα πλαίσια της πολιτικής μας, στα πλαίσια της πολιτικής ανάπτυξης ή της τράπεζας ανάπτυξης και επίσης θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερη συνέπεια, περισσότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη προβολή με αυτή την πρόταση όσον αφορά τη δράση τη Ένωση. γιατί αυτή τη στιγμή εμεί είμαστε η βασική χορηγή της βοήθεια. βοήθειας παρόλα αυτά όμω, όπω έχει σήμερα η κατάσταση δεν έχουμε την ανάλογη προβολή ούτε αποτελεσματικό επομένω τον έχουμε μια τέτοια ενωσιακή ε, κοινοτική πλατφόρμα και όλα αυτά που να μπορούμε να τα συσπηρώσουμε είναι μια ιδέα πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον Νομίζω ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα αλλά και το ότι θα ξεκινήσει η λειτουργία αυτή η υπηρεσία εξωτερική δράση τη Ένωση είναι μια ευκαιρία τόσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την αναγκαία υποστήριξη για να έχουμε αυτή την ενιαία πολιτική. Άλλα δύο τώρα σημεία για να ακούσω την ε, γνώμη σα για ε, αυτά, την τόσο αξιόλογη έκθεση τη κ. Γκουίνεθ Τζόνς που την οποία και ευχαριστούμε για όλες αυτέ τις ιδέες που μας έδωσε. Πρώτα πρώτα όσον αφορά την εκταμείευση και την, και την ανάπτυξη των κινδύνων, όσον αφορά την εκταμείευση, θέλω να σας τονίσω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά το τι γίνεται από τη μια χρονιά στην άλλη ίσως ε, πάνω στην πορεία είναι σημαντικό. Όμως είναι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι οι επιδόσεις μας δεν είναι τόσο καλές όσο αλλού σε για άλλα θεσμικά όργανα και το σημαντικό είναι για την απόδοση να δούμε ότι πρώτα πρώτα τα project της ε, ΕΤΕ, τα χρηματοδοτικά και κυρίως όσον αφορά τα project σε σχέση με τις ΜΜΕ ε, είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τον εθνικό προπολογισμού. Καλό ή κακό, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αλλά δεν, έτσι δεν έχουμε κανένα είδου γρηγορότερη ε, εκταμείευση. Χρηματοδοτούμε όχι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά μόνο τι ΜΜΕ μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των τραπεζών αυτών. Άρα προσοχή όσον αφορά το τι γίνεται με τι πιστώσει μα και τη ζήτησή του. Δεύτερο θέμα, το οποίο μα ε, αφορά εδώ είναι ότι κάποτε η, η ΕΤΕ έχει ακόμα και για ντάμπινγκ, γιατί ήμασταν λιγότερο ακριβοί από ότι τα άλλα θεσμικά ιδρύματα. Σήμερα όμως είναι το ανάποδο. Δεν είμαστε καθόλου ανταγωνιστικοί γιατί ε, όλοι έχουν κάποιο είδου επιδοτήσεις, χορηγίες και όταν έρχεται η ώρα του, του δανεισμού τότε ο, ο καθένας πάει ε, εκεί που είναι τα πιο, τα πιο φτηνά λεφτά. Τώρα, σαν αφορά του κινδύνου. Πρώτα-πρώτα εδώ το θέμα είναι τι γίνεται με το κεφάλαιο της τραπέζης, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε μια αναλογία που μας περιορίζει σε σχέση με το πόσα δάνεια δίνουμε ή πόσους κινδύνους αντιλαμβάνουμε. άρα θα πρέπει να είμαστε προσκλητικοί αν δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να μας δώσουν λεφτά. Ε, και εν πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά με την ε, Κομισιόν, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε περισσότερο, να πιάσουμε περισσότερο τόπο τα δάνεια αλλά και οι χορηγίε και κατά κάποιο τρόπο να ανακουφίσουμε την πίεση στο, στο, στο κεφάλαιό μα και έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μα καλύτερα. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και τώρα. Το, κύριο, το λόγο για περίπου 7 έχει ο κύριο Κασόνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάσω σήμερα την άποψη της Κομισιόν για την εντολή αυτή την εξωτερική. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζουμε εδώ την πρόταση Κομισιόν όπως παρουσιάστηκε στη πρώτη φορά στις 21 Απριλίου και στάλει στο Κοινοβούλιο στις αρχές αυτού του μήνα. Ε, νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση είναι ισόρροπη ε, και επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να υλοποιήσει την εξωτερική της εντολή. Η νομική βάση εκπνέει το 2011. Άρα δηλαδή ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή η συζήτηση που γίνεται στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως ήδη ανέφερε ο Ντομινίκ Κρανκούρ, η πρόταση της Επιτροπής εμπνέεται σε μεγάλο βαθμό από την εντολή Ευρώπη 2 δις. Μια πρόταση που την είχαμε εμπνευστεί κυρίως ε, για θέματα κλιματικής αλλαγής. Κατόπιν όμως ε, πρόκειψε μια σημαντική αλλαγή και θα επανέλθω σε αυτό ε, όταν θα κάνω τα σχόλια για την έκθεση της Griffith Jones. Εμείς λοιπόν προτείναμε να τροποποιηθεί να τροποποιηθούν οι περιφερειακοί στόχοι ε, που έχουν σχέση με την εντολή της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα καθοριστικό σημείο της έκθεσης ε, της ε, κυρίας Τζόνς, δηλαδή να μπορεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επεμβαίνει στις διάφορες ε, περιφέρειες με τις ίδιες ακριβώς δραστηριότητες. Κατόπιν, αποδώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο να υιοθετήσουμε την παλαιότερη συζήτηση που είχε γίνει στο Κοινοβούλιο και την τρέχουσα νομική βάση όπου το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, πρέπει ε, να ταχθεί περισσότερο υπέρ ε, της χορήγησης πιστώσεων. Όπως είπε και ο συναδελφός μου, αυτό προϋποθέτει την σταδιακή αύξηση και ένταση των προσπαθειών ελέγχου της, ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων. Άρα δηλαδή ε, χρειάζεται περισσότερο προσωπικό για να υλοποιήσει όλους αυτούς τους στόχους. Το θέμα δεν είναι να δώσει κανείς ε, μόνο εντολή στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αν δεν έχει τους πόρους να τα κάνει όλα αυτά. Το ανθρωπινό δυναμικό κυρίως και εδώ η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καθοριστική σημασία. Αυτό το θέμα της ε, ανάπτυξης για μας είναι σημαντικό. Πιστεύουμε ότι εκεί μπορούν ακόμα να γίνουν πολλά πράγματα και προτείνουμε την σταδιακή ε, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στους κοινωνικού τομείς όπως είναι η παιδεία παραδείγματος χάρη. Αυτό πάλι είναι ένα θέμα ε, το οποίο αναφέρεται στην έκθεση της κυρίας Γκριφίδ. Ένα άλλο πράγμα αφορά σε κάτι που εμείς είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο. Πρόκειται για το θέμα ε, των κριτηρίων ανάπτυξης. Δηλαδή, όταν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εξετάσει περισσότερο τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, ε, για να, τα, για να πετύχουμε το στόχο μας ε, πρέπει να δούμε, να εξετάσουμε καλύτερα τις, ε, τους μηχανισμούς ε, δανειοδότησης. Το τελευταίο που θέλω να πω στην πρότασή μας έχει σχέση με την ε, ανάγκη αντί να μεταφραστούν σε περιφερειακό επίπεδο αυτοί οι υψηλοί στόχοι και να εξετάζει κανείς το πώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να καταρτίζει περισσότερα έγγραφα με τη μορφή των ε, περιφερειακών οδηγιών. Μετά βέβαια από παρεμβάσεις ε, του Συμβουλίου και της ε, Κομισιόν στην έκθεση Καντεσούρ δεν αναφέρεται, αλλά αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής. Πρόκειται εδώ για την επέκταση της ε, γεωγραφικής ε, εμβέλειας ε, της εντολής και αναφέρονται προϋποθέσεις απέναντι στην Ισλανδία, την Λευκορωσία, το Ιράκ, την Καμπότζη. Εκεί λοιπόν θα θέλαμε να υπάρχει διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, κατά τη διάρκεια της έγκρισης της εντολής. Επιτρέψτε μου να κάνω και κάποια άλλα σχόλια που αφορούν σε αυτή την πολύ καλή έκθεση και να ευχαριστήσω όχι μόνο την καθηγήτρια κυρία Τζόνς αλλά και τον κύριο Μπέρμαν γιατί επέτρεψαν στην Κομισιόν να παρέμβουν στην ομάδα εργασίας ε, προετοιμασίας αυτής της έκθεσης που είναι πάρα πολύ καλή και προσφέρει τροφή για σκέψη. Ε, αυτό που είναι σημαντικό είναι να κατανοήσει κανείς ότι τώρα η τράπεζά μας ε, λειτουργεί μετά από εντολή του Συμβουλίου ε, και του Κοινοβουλίου. Εσείς δηλαδή είσαστε εκείνοι που αποφασίζετε για τις εξωτερικές δράσεις της ε, Τράπεζας Επενδύσεων. Δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμεθα για το ότι δεν είναι παρούσα η ε, Τράπεζα Επενδύσεων σε όλες τις χώρες, γιατί αυτό πρέπει να ξεκινήσει εδώ από μια κοινοβουλευτική συζήτηση. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι εγώ προσωπικά συμμερίζομαι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ακόμα μεγάλο περιθώριο για να αναλάβει κινδύνους και σε εξωτερικό επίπεδο. Η ε, τράπεζα έχει ισοσκελισμένους ε, ισολογισμούς και η ύπαρξη εγγύησεων νομίζω ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτό έτσι ώστε η Τράπεζα Επενδύσεων να μπορεί να εστιάσει την προσοχή της ακόμα και σε επικίνδυνες χώρες. Και βεβαίως να γίνονται και επενδύσεις ε, σε χώρες πιο ασφαλείς. Νομίζω λοιπόν η Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να αναπτύξει περισσότερες δραστηριότητες και στους δύο τομείς. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να πω ότι ο ευρωπαϊκός ε, προϋπολογισμός, ο εξωτερικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή ε, χρησιμοποιείται περιορισμένα. Δεν νομίζω ότι ξεπερνά το 3-4% ε, της γραμμής για εξωτερικές δραστηριότητες. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική μόχλευση στις δραστηριότητες της Επιτροπής ε, και στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα θέλαμε να υπάρχει μια σταδιακή αύξηση, ίσως περίπου στο 10%. Ε, αυτό θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Και παράλληλα ε, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε έναν προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι περιορισμένος. Θα υπάρχουν περιορισμοί στα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά με την επόμενη δημοσιονομική πειθαρχία. πειθαρχία. Πάνω θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε έναν περιορισμένο προεπλογισμό και την ανάγκη χορήγησης δανείων. Το τελευταίο που θέλω να αναφέρω και ίσως και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει αυτό το θέμα της ε, εποπτείας από πλευράς Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι αυτό είναι ε, μια καινοτομία στη συζήτηση που γίνεται για την εντολή. Στην τελευταία συζήτηση πριν από τον Ιούλιο του 2009 όταν εγκρίθηκε η νομική βάση ε, στόχος ήταν να επανέλθει η νομική βάση. Ε, τώρα λοιπόν ε, θέλουμε να ξανασυζητήσουμε για την νομική βάση του Κοινοβούλου και με μεγάλη μας χαρά θα ακούσουμε τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ και το λόγο τώρα έχουν οι βουλευτέ Αν υπάρχουν κάποιε ερωτήσει που θέλετε να θέσετε. Κύριε Γερέρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα συγχαρητήρια προ ε, τον εισηγητή. Τον κύριο Τάις γιατί πρόκειται για πάρα πολύ περιεκτική έκθεση, αναλυτική, ε, διότι βλέπουμε πόσο συναρπαστικό ε, είναι ο εισηγητή. Άλλωστε είναι συναρπαστική προσωπικότητα, πολύ ενδιαφέρουσα και αυτό κάνει πάρα πολύ και στην παρουσία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θα πρέπει να σα πω ότι εδώ διάφοροι συνάδελφοι στην Επιτροπή μα και γενικότερα η Επιτροπή μα ήδη έχουμε διαφοροποιημένε ο καθένα ε, σχέσει μέσα στο Κοινοβούλιο ή τέλο πάντων και εκτό Κοινοβουλίου σε σχέση με την ΕΤΕ. Τούτο καταδεικνύει πόσο Ενδιαφέρουσα είναι για μας η δραστηριότητα της τράπεζας. Αλλά και το τι διαφορετικές προοπτικές βλέπει ο καθένας. Επομένως να δούμε τι μέλλον έχει ε, η πολιτική της ανάπτυξης σε σχέση με τις δραστηριότητες της τράπεζας. Ο κύριο Ρένο, ο επίτροπο ε, που έχει το χαρτοφυλάκι των οικονομικών θεμάτων, πρόσφατα λέγω που μα είπε ότι θα πρέπει η τράπεζα να τονίσει περισσότερο, να προσέξει περισσότερο την πολιτική τη ανάπτυξη. Και πιο συγκεκριμένα μας είπε για κάποιου είδους προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με την περιβαλλοντική υποδομή, με τη μεταφορά υδάτων, με κάποιο είδους βιώσιμη πολιτική μεταφορών, υγεία αλλά και παιδεία. Ταυτόχρονα δε η Επιτροπή Σοφών ανέλησε την ε, μεσοπρόθεσμη μεταρρύθμιση της ε, ΕΤΕ. Και εκεί επίσης στο κείμενό τους ε, επισημάνθηκε ότι στα πλαίσια αυτού του προφίλ της ε, τράπεζας θα πρέπει ε, να προσεχθεί περισσότερο η εξωτερική δράση της ε, τράπεζας. Γιατί θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι ακόμα ένα μέσο άσκηση εξωτερικής πολιτικής από την Ένωση. Και επομένως θα πρέπει στην πλατφόρμα που είπαμε, στην πλατφόρμα που θα φτιαχτεί, να μπορέσουμε να έχουμε την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, να τη συγκεράσουμε με την εξωτερική δράση της τράπεζας ε, και έτσι να υπάρχουν καινούργιες δεσμοί, καινούργιες σχέσεις με, τις, με κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης. Επομένως, έτσι αναπτυχθεί μια πολιτική η οποία όλο και περισσότερο να προσέχει την αναπτυξιακή συνεργασία. Σε αυτή την έκθεση, διότι όσον αφορά τι επιπτώσει τη κρίση, για τις αναπτυσσόμενες χώρες, είχα την ευκαιρία να είμαι ο συγητής. Και είπαμε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναλάβει δράση και δραστηριότητα να αναπτύξει για κάτι που είχε τονιστεί. Ότι δηλαδή θα πρέπει οι εγγύσεις, οι επενδύσεις, οι δραστηριότητες της ΕΤΕ να μην γίνονται μέσω φορολογικών παραδείσων, ούτε να γίνονται κατά κάποιο τρόπο έμεσα. Θα πρέπει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αυστηρότητα και σοβαρότητα να δούμε τι θα κάνει η τράπεζα σε αυτόν τον τομέα, σε αυτές τις δραστηριότητε. Και νομίζω δε ότι είμαστε εις θέση να φροντίσουμε σε αυτήν την μεσοπρόθεσμη μεταρρύθμιση, αναθεώρηση του ρόλου της ΕΤΕ και στο τι θα γίνει με το μέλλον της, να δούμε πώς μια τέτοια προσωπικότητα της Ένωσης να προβληθεί. Αυτό σας θέτω σήμερα ως ζήτημα. Να δούμε πώς θα επανακαθοριστεί το προφίλ της τράπεζας, χωρίς να αρνηθούμε το παρελθόν της. Όμως θα πρέπει να ενισχυθεί η πτυχή ανάπτυξη ε, Επομένω, και εμείς θα πρέπει με τη σειρά μας να τους στηρίξουμε ε, όλο το Κοινοβούλιο και βέβαια πιο συγκεκριμένα η δική μας Επιτροπή. Ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Γκέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο προλαλή σα, πάρα πολύ αυτό θα τα είπε όσον αφορά τους επένους που αξίζουν στον ε, εισηγητή. Και επομένω τα είπε τόσο καλά που δεν μπορώ να βρω καλύτερα λόγια για να επενέσω τον συνάδελφο και φίλο. Δεύτερον, διακομματική είναι η συνεργασία μας σε αυτή την Επιτροπή. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχουν κομματικά συμφέροντα. Τώρα, όσον αφορά αυτά τα οποία είπε η Κομισιόν, γενικά συμφωνώ, θα πρέπει εκεί πέρα να μην έχουμε καμία δυσκολία να δανείσουμε, θα πρέπει να ε, υπάρχουν ε, κάποιες χορηγίες, κάποιοι δανεισμοί ή δάλλως ε, εάν δεν πληρούνται κάποιες υποθέσεις δεν είναι δυνατόν η ΕΤΕ να, να, να, να δανείζει και άρα δεν μπορούμε να την, να την κατηγορούμε ότι δεν δανείζει αρκετά. 20-30% 40 χρόνια λέμε για 40 δις δολάρια τα οποία ματιώνονται ως δάνεια για κάποιους βάσιμους λόγους. Οπότε γι' αυτό και τώρα θέλω να ρωτήσω ε, στους συναδέλφους της ΕΤΕ αλλά και της ε, Κομισιόν να μας πούνε τι γίνεται όσον αφορά αυτή τη συνέργεια μεταξύ της Κομισιόν και της ε, ΕΤΕ. Τι γίνεται. Είναι δυνατόν να έχουμε συγκεκριμένη έκφραση αυτή της ενέργειας στα πλαίσια της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχει ωφεληθεί όλη η Αφρική από τα δάνεια. Όμως, μήπως πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποια στρατηγικά προγράμματα, ιδίως όσον αφορά τις εναλλακτικέ ενέργειες, για παράδειγμα. Ναι, πώς μπορούμε να είμαστε φιλόδοξοι. Να έχουμε όμως κάποια προγράμματα ευρεία κλίμακα. Τώρα όσον αφορά αυτά τα ποσά, τα 7 δις που είπε η Κοπεχάγη όσον αφορά την, την, την, την, την κατανομή του, συγγνώμη, 2010-2012. Μπα και θα πρέπει αυτά τα, να τα χρήματα τα ρίξουμε σε κάποια μεγάλα προγράμματα τα οποία θα συγκεντρώνουν τη συνεργασία δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Α πούμε αυτά τα joint ventures βορρά-νότου. και να ωφεληθούν ακόμα και οι χώρε του Βορρά. Να ωφεληθούν από αυτά τα δάνεια τη. ΕΤΕ. Αλλιώς, εσαΐ θα συζητάμε τα ίδια πράγματα χωρίς να έχουμε κανένα αποτέλεσμα αυτό. Επίσης, για να μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτή τη διακυβέρνηση, ίσως θα πρέπει να έχουμε να βάλουμε ως όρες αντισόμενες χώρες τη βελτίωση της διακυβέρνησης. Και κατά αυτόν τον τρόπο να εξασφαλιστούν τα ποσά αυτά, τα, τα ποσά τα οποία προέρχονται από τις βιομηχανικές χώρες. Ίσως με τέτοιου είδους στρατηγική θα μπορούσαμε να τονώσουμε κάπως παραπάνω την, ε, τη συνεργασία δημοσιοδητικού τομέα. Γιατί τα βήματα πρόοδου σε αυτό το τομέα είναι πάρα πάρα πολύ μικρά. Έχουμε γι' αυτό το African Business Forum εδώ και ε, κάποια χρόνια. Λειτουργεί αλλά δεν βαδίζει, δεν προχωράει. Δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ λοιπόν. Και τώρα δώσουμε για πάλι το λόγο ή στον κύριο Κρενικούρ και στον κύριο Κασόνια και κατόπιν θα ξαναλάβει τον κύριο Μπέρμαν. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα ε, θα προσπαθήσω να τοποθετηθώ ε, σε αυτά ε, που είπαν οι κύριοι Κεραίρο και Γκέρονς. Πράγματι, αυτή η ιδέα της πλατφόρμας, όπως ακριβώς την περιγράφει η έκθεση του εισηγητή, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με την έννοια ότι θέλουμε να υπάρχει οικονομική υποστήριξη στις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να δώσω και μία απάντηση και στον κύριο Γκέρινγκ, ξέρετε αυτό είναι το είδος πλαισίου που έχουμε κατά νου για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, κλιματικής αλλαγής. Οι ε, προκλήσεις μετά την Κοπεχάγη είναι τεράστιες κυρίως οι μακροχρόνιες. Εμείς λοιπόν έχουμε καταθέσει μία πρόταση να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έννοια της ε, πλατφόρμας έτσι ώστε να, ε, να υποτάξουμε όλες ε, τις τους που μπορούν να υπάρχουν κάτω από τη ΣΜΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. με αυτόν τον τρόπο επιθυμούμε να προσεγγίσουμε το όλο θέμα. Και αυτό ισχύει και για μεγάλα και για μικρά προγράμματα. Γιατί νομίζω και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Ε, τώρα όσον αφορά τα οικονομικά κέντρα τα οποία ανέφερε ο κ. Γκερέρο, πρέπει να είστε σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το θέμα αυτό το λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά. Ε, δεν πρόκειται πάντα για ένα εύκολο θέμα. Ε, Παρ' όλα αυτά εμείς ε, είμαστε πολύ πιο μπροστά από οποιονδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Αυτή τη στιγμή ε, δαπανάμε πολλά χρήματα για να πείσουμε άλλους οργανισμούς να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο που βρισκόμαστε και εμείς. Γιατί δεν έχει νόημα να ε, λέμε σε μία χώρα ή σε ένα επενδυτικό φορέα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ε, και ότι είμαστε αναγκασμένοι να πάμε από το ένα φορέα στον άλλο. Πρέπει παντού να υπάρχει η ίδια προσέγγιση. Κάτι που ξέρετε πάρα πολύ καλά κύριε Πρόεδρε είναι το θέμα του να καταρτιστεί ένας κοινό κατάλογος χωρών. Και δυστυχώς αυτό ξεφεύγει από τις ικανότητες μιας τράπεζας όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να περισσότερο στην Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να αποφασίσουν για το θέμα σε πολιτικό επίπεδο. Τέλος, όσον αφορά τι ε, υπερχρεωμένες ε, χώρε και την ανάγκη ε, να υπάρχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Τράπεζα. Θέλω να σας πω ότι εμείς καθυστερήσαμε εδώ λιγάκι γιατί ήμασταν σε μία ε, συνάντηση με την Κομισιόν όπου εξετάζαμε ακριβώς αυτό το θέμα. Ε, για να σημειώσουμε και επιτύχουμε πρόοδο σε αυτό το θέμα το οποίο το επιθυμούν όλοι οι μέτοχοι. Ευχαριστούμε πρόεδρε και Ντομινίκη γιατί είπες ε, τα περισσότερα από αυτά που θα ήθελα να πω. Όσον αφορά σε αυτό το θέμα ε, επί το οποίο αρχίζουμε τώρα να σκεπτόμεθα το θέμα της ε, πλατφόρμας έτσι ώστε με πιο έξυπνο τρόπεζο να μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις της Κομισιόν και τους άλλους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ε, βεβαίως ε, μας ενδιαφέρει και η διμερής ε, συνεργασία με πολλές τράπεζες. Όσον αφορά τώρα στο θέμα του να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε, να διασπείρουμε τους πόρους σε διάφορα προγράμματα, εγώ θέλω να σας πω ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τις απόψεις του κυρίου Γκέρονης. γιατί ακριβώς αυτό θέλουμε να κάνουμε μέσα από τις ε, κατευθυντήριες ε, γραμμές, κυρίως μέσα από την εντολή ε, για την κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα εξτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το εξτάσουμε με στρατηγικό τρόπο. Εγώ λοιπόν ε, θα ήθελα με μεγάλη μου χαρά να ακούσω περισσότερες απόψεις για αυτά που μας είπατε ε, όχι μόνο τα προγράμματα στα οποία ε, θα πρέπει να κατευθύνεται η εντολή, αλλά και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτούς τους τομείς. Όσον αφορά τις υπερχρεωμένες χώρες, συμφωνώ εδώ με τον Ντομινίκ, μέσα από την εγγύηση επενδύουν οι περισσότερε χώρε, αλλά και χωρί την εγγύηση το επίπεδο μόχλευση σε ορισμένε χώρε είναι τέτοιο που δεν είναι εύκολο κανεί να επέμβει. Και δεν μπορεί κανεί ε, να προσφέρει νέε επενδύσει όπω αυτέ, να εγγύσει με συγχωρείτε όπως αυτές που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι πώ μπορούμε να συγκεντρώσουμε του πόρου ε, και από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να υπάρχει ε, και η απαραίτητη κάλυψη αυτών των δανεισμών. Ευχαριστούμε κύριε Μπέρμαν, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε. Τώρα να σας το πω στα γαλλικά. Όσον αφορά αυτή την, όπως είπατε, ε, αυτά τα οποία είπε ο ο εξαίρετος συνάδελφος ο κύριος ε, πάλι καλά που εδώ πέρα ανταλλάσσουμε ε, ε, τις φιλοφρονίες γιατί αυτό δεν συμβαίνει έξω από το κοινοβούλιο. Πολύ σπάνιο. Τέλος πάντων. Να αναφερθώ σε κάποια τα οποία δεν μπόρεσα να σας τα θίξω όσον αφορά την ε, έκθεση Wynne Jones. νομίζω ότι έχει διαμορφωθεί κάποια συνένεση που, αυτό αντικατευθύνεται και στην έκθεση των σοφών και στην έκθεση της Κομισιόν και στην ε, έκθεση της Γκούνις Τζόνς. ότι δηλαδή είναι φανερό ότι αυτό το οποίο χρειάζεται η τράπεζα να καταστεί ένα εργαλείο χρήσιμο για την ανάπτυξη. Δεν είναι δυνατόν να, να, να, να υπάρχουν μόνο αυτού του είδους οι επιδοτήσεις. Χρειάζεται ένα τραπεζικό εργαλείο πολιτικής, δημόσιο. Πάει αυτό. Μία τράπεζα η οποία να ασχολείται όχι μόνο με αυτά που ασχολείται στο παρελθόν, δηλαδή επενδύσεις σε, σε υποδομές, βιώσιμης ενεργικής πολιτικής, σε ΜΜΕ, σε δραστηριότητες μέσα στην Ευρώπη παρά έξω. Τώρα χρειάζεται κάτι καινούριο. Και αυτό να γίνεται υπό όρους και προϋποθέσεις κάποιας ανάπτυξης βιώσιμης, με διαφάνεια δηλαδή να μην χρησιμοποιούμε αυτές τις υπεράκτιες εταιρείε, offshore, φορολογικούς παράδεισους. Και δεν το λέω αυτό μόνο επειδή το είπε και η πρόεδρός μας, η Ζολή. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ολοφάνερο και μόνο θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία ακόμα πιο στενή με τα κράτη-μέλη. FMO, ΚΑΒ και λοιπά, με τους εθνικούς φορείς σαν εταιρείε και επίσης να υπάρχει μια προστευμένη εντολή ούτω ώστε να υπάρχει μια εντολή που να μπορεί να καλύψει όλες τις περιοχές και περιφέρειες ούτω ώστε να υπάρχουν κάποιε αποστευμένες διαδικασίε γιατί ένα κομμάτι της βραδύτητας της ε, ΕΤΕ είναι στο ότι έχουμε κάποιε διαδικασίε εκεί υπερβολικά περίπλογε. Επιδέχονται απλούστευση, σίγουρα. Και επίση θα πρέπει και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή πρόταση αυτή της Κομισιόν και της Επιτροπής των Σοφών να χρησιμοποιηθούν τις, αυτά τα της προαιρετικής ε, εντολής, τα δύο εκατοδείς να χρησιμοποιηθούν αυτά τα οποία αφορούν το κλίμα να χρησιμοποιηθούν. Και το λέει και η Gwyneth Τζόν, την έκθεση. Πάρα πολύ καλά όλα αυτά, αλλά αν θέλουμε να έχουμε μια κρατική δημόσια τράπεζα που να παίζει το ρόλο της στο, στο, στην προσπάθεια για ανάπτυξη θα πρέπει αυτή η τράπεζα να βοηθάει αυτές τις χώρες να μπορούν επομένω όλοι να έχουν ε, πρόσβαση ε, σε αυτά τα κεφάλαια που το οποίο δεν ισχύει σήμερα. Θέλει δηλαδή ο Γιώργος να βρει ένα φορτηγάκι να μπορεί να πάει λίγο παραπέρα τα ζώα του να τα πουλήσει και αυτό ισχύει ακόμα και σε κάποια γυναίκα που θέλει μια ραπτομηχανή να φτιάξει ένα γραφείο που είναι τώρα μικρό να το κάνει λίγο πιο μεγάλο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη ε, των ε, αναπτυσσόμενων χωρών και είναι κάτι το οποίο θα μας ωφελήσει όλους. Ευχαριστώ, και πάμε στο 7ο σημείο Όπως ξέρετε σχετικά με το δικαίωμα εξετάσεως των ε, εγγράφων προγραμματισμού ε, για την νομοθεσία από πλευράς ε, αναπτύξεως. Όπως ξέρετε έχουμε λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένα έγγραφα στρατηγικά και θα παρακαλούσα τώρα τις ομάδες εργασίας να παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους. Ο κύριος Νόισερ έχει την, την εκπροσώπηση της ομάδος Α και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είμαι ο μόνος από την ομάδα εργασίας Α για να παρουσιάσω την έκθεσή μου Είχαμε ε, ανταλλαγές απόψεως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σχετικά με τα στρατηγικά έγγραφα για το Βιετνάμ, την Μαλαισία, τη Βιρμανία και την Καμπότζη στις 28 Απριλίου και ξανασυζητήσαμε την Καμπότζη και στις 5 Μαΐου. Καταρχήν όσον αφορά το Βιετνάμ. Η ομάδα εργασίας Α θεωρούν ότι ε, υπάρχουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα, καταρχήν η υγεία, ε, και ε, μέχρι στιγμής οι προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει, θα έπρεπε να υπάρξει βελτίωση Επίσης ε, ε, θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες στο μέλλον και ε, να διευκρινίσουμε το θέμα της επιλεξιμότητος όσον αφορά την διακυβέρνηση και τον διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της χώρας. Όσον αφορά την Καμπότζη μπορεί να δοθεί βοήθεια αλλά δεν υπάρχει μεγάλη διαφάνεια και έχουμε ακόμη πολλά να πάνε τα ερωτηματοκιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχεται ότι όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση και την αναθεώρηση υπάρχει ακόμη εγγενής διαφθορά και δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί σχετικοί νόμοι. Θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συζήτηση με την κυβέρνηση και άλλους ενδιαφερόμενους πόσο θα μπορέσει να αποδώσει περισσότερο το πρόγραμμα αυτό και ε, γι' αυτό αναφέρεται ότι ε, τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων ε, πρέπει να αποδίδουν και πρέπει να προϋποτίθεται ότι υπάρχει και διαφάνεια και απολογισμός. Χρειάζονται τακτικές εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη των δικτών και ε, να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο το οποίο να εξαρτάται από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων εκλεξιμότητος προτού υπάρξει οποιαδήποτε εκταμίευση. Όσον αφορά τώρα τη Μαλαισία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ασχοληθεί περισσότερο με τα εξή θέματα. Πρώτον, ε, το δικαίωμα των ε, ε, ηθαγενών σε ορισμένα μέρη της χώρας θα έπρεπε να βελτιωθεί η, ε, η κατάσταση από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδίως όσον αφορά τις ελευθερίες και ε, ο στόχος της χιλιετηρίδος παριθμών 6 θα έπρεπε να επιτευχθεί μέχρι το 2015. Εν ονόματι του κυρίου Κασμάρεκ θα μπορούσα επίσης να παρουσιάσω την έκθεση της Βυρμανίας και ε, να σας πω ότι θα πρέπει ε, να ληφθούν ε, υπόψη οι ε, λεπτομέρειες της πολιτικής καταστάσεως και οι μελλοντικές δυνατότητες για να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην συγκεκριμένη χώρα. Επίσης θα έπρεπε να διοχετευθεί το θέμα των ε, φύλων ή ε, της ισότητας των φύλων ή την έκθεση και θα έπρεπε να υπάρξει ε, συγκεκριμένο πλαίσιο για τη βοήθεια προς τη χώρα. Τώρα όσον αφορά η κυρία Κρετού ε, για την επόμενη έκθεση ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δώσει στο Κοινοβούλιο περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική κατάσταση και όσον αφορά την φάση εφαρμογής θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε ότι η οικονομική ε, βοήθεια ε, εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε το, οι στόχοι της DCI να εφαρμόζονται ιδίως όσον αφορά την ε, εξάλληψη της στόχιας και τα συμπεράσματα είναι ότι σε αυτή τη φάση της διεργασίας βάσει ε, των εγγράφων η ομάδα εργασίως Α ε, προτείνει να μην υπάρξει αναθεώρηση στα έγγραφα ε, των χωρών αυτών βάσει της επιτροπολογίας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 35 της DCI και να θεωρήσουμε ότι έχει εκπνεύσει προθεσμία για το δικαίωμα εξετάσεως. Θα πρέπει να προωθηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συγκεκριμένα ερωτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διατύπωση του σχετικού ετησίου προγράμματος και να υπάρξει μία ε, αναθεωρημένη μορφή των εγγράφων όσον αφορά την Βυρμανία, την Μαλαισία, το Βιετνάμ και την ε, Βυρμανία και θα τα λάβει υπόψη της. Ευχαριστώ συμφωνούν ε, τα μέλη της Επιτροπής με τα πορίσματα που αναγνώστηκαν για την ε, πρώτη ομάδα εργασίας. Τότε θεωρώ ότι ε, έχει ολοκληρωθεί το δικαίωμα δημοκρατικής εξετάσεως για αυτά τα σημαντικά έγγραφα και κλείνω τη διαδικασία. Δίνω τώρα τον λόγο στην κυρία Λέβιν ή στον κύριο Ντεβά για την ομάδα εργασίας Β για να μας παρουσιάσει τους στόχους αυτής της ομάδας εργασίας. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εμείς ε, στην ομάδα εργασίας Β εξετάσαμε την ε, ενδιάμεση έκθεση για την Ινδία, τον Νεπάλ και το Πακιστάν και ε, παρουσιάσαμε τα ε, συμπεράσματά μας. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την Ινδία. Η Ινδία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, έχει το ενέκτο του παγκόσμιου πληθυσμού και δυστυχώς και το 1 τρίτο των φτωχών του κόσμου. Η χρηματοδότηση μέσα από το πολιετές πρόγραμμα ε, κατακαιρματίζεται, σε, σε δύο τομείς προτεραιότητες. Οι δράσεις στο πρώτο τμήμα αφορούν την υποστήριξη του κοινωνικού τομέα, κυρίως της υγείας και της παιδείας. Αυτές οι προτεραιότητες ε, έχουν ως στόχο τα προγράμματα μεταρρύθμισης και επίσης έχουν και ως στόχο να επιτύχουν κάποια πρόοδο, γι' αυτό η προτεραιότητα υπαριθμών 1 είναι σημαντική. Η προτεραιότητα υπαριθμών 2 αφορά την κοινωνία των πολιτών, ε, τον πολιτισμό και τους ακαδημαϊκούς τομείς. Και εκεί προβλέπεται και ο διάλογος ε, με τις διάφορες ρέσεις και ε, προβλέπονται επίσης και ακαδημαϊκές ανταλλαγές διαπιστώσαμε ότι η δεύτερη προτεραιότητα δεν έχετε άμεση σχέση με την ε, καταπολέμηση της φτώχειας. Μάλιστα, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δεν δείχνουν και μεγάλο ενθουσιασμό για αυτή την προτεραιότητα. Από το 2007 έως το 2010 η προτεραιότητα υπαριθμών 1 πήρε το 70% των κονδυλίων και η υπαριθμών 2 προτεραιότητα ε, το 30%. Πιστεύουμε ότι το πολιτές πρόγραμμα για την Ινδία από το 11 έως το 13 θα πρέπει να εστιάζει περισσότερο την προσοχή του στην ε, προτεραιότητα υπαριθμών 1. Η πρόταση της Κομισιόν αναγνωρίζει βέβαια αυτό το γεγονός. όλα αυτά, τα στοιχεία που έδωσε η Κομισιόν αφήνουν περιθώριο ε, να έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Από το 11 μέχρι το 13 μιλάμε για το 70 μέχρι το 85% προτεραιότητα 1, δηλαδή παιδεία και υγεία και 15 μέχρι 30% για την ε, προτεραιότητα υπεριθμών 2. Άρα ε, δηλαδή μπορεί να μην υπάρχει καμία αύξηση στην προτεραιότητα υπαριθμών 1. Και αυτό είναι παντελώς ε, απαράδεκτο. Επίσης ε, έχουμε και κάποιες εμφωλίες όσον αφορά το Erasmus Μούντις. Είναι απολύτως απαραίτητο να μην χορηγηθεί βοήθεια με τη μορφή των υποτροφιών για τους Ευρωπαίους φοιτητές και καθηγητές. Εξάλλου το Erasmus Mundus ε, μπορεί να συμβάλλει ε, στην ε, αφέμαξη, στην ροή των εγκεφάλων. Εάν λοιπόν αυτό το πρόγραμμα πρόκειται να συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη της Ινδίας, η επιλεξιμότητα είναι πολύ σημαντική και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί για την Ινδία. Πώς μπορεί κανείς να πιέσει τους ανθρώπους να επανέλθουν εάν δεν το επιθυμούν. Όσον αφορά την ε, συμμετοχή ε, διαφόρων άλλων ενδιαφερομένων. Το Κοινοβούλιο δεν εισακούεται για την ενδιάμεση έκθεση. Εμείς λοιπόν προτείνουμε να μην απορριφθεί η έκθεση για την Ινδία υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουμε ικανοποιητικέ απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μέχρι τις 21 Μαΐου για δύο βασικά θέματα. Πρώτον, η Επιτροπή μπορεί να εγγυηθεί ότι θα υπάρχει σημαντική αύξηση όσον αφορά τα κονδύλια που χορηγούνται για την προτεραιότητα υπαριθμών 1. Τουλάχιστον το 80% των κονδυλίων ε, αυτό αφορά. Μετά, μπορούμε να εισάγουμε την επιλεξιμότητα στο ο βίντους Μούντις για να αποφύγουμε την διαρροή των εγκεφάλων και έτσι ώστε οι ερευνητές και φοιτές πραγματικά να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας τους. Κατόπιν, όσον αφορά τον ΠΑΛ, η ομάδα εργασίας είναι ικανοποιημένη. Η, ε, ο γενικός προσανατολισμός επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της ε, αναθεώρησης και οι τρεις τομείς προτεραιοτήτων παρέμειναν οι ίδιοι. Ε, σταθερότητα και ειρήνη, ε, εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη. Όπως θα θυμάστε κυρία Πρόεδρε, υπήρξαν αναταραχές στο Καταμούντου την περασμένη εβδομάδα και τα προγράμματα της σταθερότητας είναι πολύ σημαντικά ε, καθώς καταβάλλονται προσπάθειες για να ανατραπεί η κυβέρνηση. Εξάλλου, ο προϋπολογισμός παραμένει στα 60 δις ευρώ για την περίοδο 11 έως 13. Όμως, ε, ε, στα χαρτιά υπάρχει παραδοχή ότι πράγματι υπάρχει και κάποια πρόοδος. Η πρόοδος αυτή αφορά στην ανάγκη για καλύτερη προσαρμογή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ισχύοντα συστήματα για την ενίσχυση της ε, ε, πορείας. Τα περισσότερα προγράμματα αφορούν από το 11 μέχρι το 13 και αυτά ταιριάζουν με τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί. Όμως έλεγχος θα πρέπει να γίνει στα υπόλοιπα προγράμματα τα οποία υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το στοιχείο της σταθερότητας η ενδιάμεση διαδικασία διεξάγεται ε, από κοινού ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλούς άλλους φορείς και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο διάλογος έχει λάβει χώρα στις 18 Ιουνίου του 2009 με εκπροσώπους του Κοινοβουλίου του Νεπάλ. Και έτσι λοιπόν προτείνουμε να μην υπάρξουν αντιδράσεις όσον αφορά την έκθεση για το Νεπάλ. Όσον αφορά το Πακιστάν,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 ε, θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς την κατάσταση όσο έχει και να την αξιολογήσει σωστά διότι η χρηματοδότηση αυξήθηκε από 200 εκατομμύρια για το 2008 μέχρι 2010 σε 225 για το 2011 μέχρι 2013. Ε, και εντοπιζόμαστε στον πρώτο τομέα δηλαδή ανάπτυξη της υπαίθρου και κοινωνική θετική εξέλιξη ενώ όσον αφορά τον δεύτερο τομέα την ε, παιδεία αυξήθηκε ε, σε αντιπαράθεση με το πρώτο. Ε, επίσης υπάρχει ένα θέμα ξεπλήματος βρώμικου χρήματος που είχε ληφθεί υπόψη το 2007 ε, και ε, θεωρούμε ότι έχει διευκρινιστεί και τώρα παραμένει άλλοι τομείς όπως η ανάπτυξη της υπαίθρου με μία ρήτρα ευελιξίας που θα επιτρέψει να ε, επέμβουμε σε άλλες ε, περιοχές της χώρας αν δεν μπορούμε να επέμβουμε στο βορειοδυτικό ε, τμήμα διότι όπως ξέρετε ότι υπάρχει μία περίοδος διαμαχών και ασταθείας σε αυτή την περιοχή. Επίσης τα περισσότερα προγράμματα από το 11 έως το 13 συνάδουν με τα κριτήρια αλλά θα πρέπει να γίνει προσπάθεια όσον αφορά τα προγράμματα δικαιοσύνης και προωθήσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στους σωστής διακυβέρνησης. Διότι ναι μεν όλα τα θέματα αυτά έχουν σχέση με το MDG αλλά είναι δύσκολο να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε όλα τα στοιχεία μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας. Φαίνεται ότι υπάρχουν, ε, υπήρξε μία πολύ εις βάθος εξέταση και δεν αναφέρεται όμως ε, η συνεργασία με το τοπικό κοινοβούλιο παρόλες τις προσπάθειες και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προχωρήσει αυτούς τους στόχους. Εμείς λοιπόν ε, θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε ε, κανείς να αντιλέξει την πρόθεση του προγράμματος στηρίξεως του Πακιστάν. Τώρα θα παρακαλούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας σχολιάσει σχολιάσει τα προγράμματα αυτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα καταρχήν να κάνω μερικά γενικά σχόλια. Καταρχήν, ε, χαιρετίζουμε τη συζήτηση η οποία γίνεται σε αυτές τις ομάδες εργασίας για την ε, καλύτερη ε, κατανόηση των ανησυχιών του Κοινοβουλίου και γι' αυτό θεωρούμε ότι ε, με αυτό το πρέμα θα πρέπει να καταρτιστούν τα προγράμματα. Ε, επίσης θα ήθελα να πω ότι ε, πρέπει να υπάρχει στήριξη του προϋπολογισμού και να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα θέματα αυτά διότι η τελική επιλογή γίνεται στο ετήσιο πρόγραμμα ε, ε, δράσεως και ε, σε αυτήν την τελική φάση θα περιλάβουμε όλα τα σχόλια του Κοινοβουλίου. Ενδέχεται να υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα το οποίο είναι πιο περίπλοκο όσον αφορά την βοήθεια σε χώρες μέσου προς υψηλού εισοδήματος αλλά είμαι ούτως ή άλλως ευγνώμων για την εργασία που έγινε στο Κοινοβούλιο και για τα σχόλιά τους. Οι ε, κύριοι ευρωβουλευτές έχουν πρόβλημα με την παρουσίαση η οποία έγινε αν όχι, θεωρώ ότι υιοθετήθηκαν οι αποφάσεις αυτές από την ε, Επιτροπή ε, Αναπτύξεως και ολοκληρώσαμε την δημοκρατική διαδικασία εξετάσεως των εξελίξεων σε αυτές τις χώρες. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Γκερέρο για την ομάδα εργασίας ε, ΓΑΜΑ. Εν Ευχαριστώ Πρόεδρε θα ήθελα να ε, παρουσιάσω την έκθεση αυτής της ομάδας ε, για τη στρατηγική του το Σαλβατόρ. Μετά ε, τον Μάρτιο του 2009 είχαμε την ευκαιρία για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας να αναλάβει την εξουσία ο πρόεδρος Φούνες, ο οποίος τώρα πλέον αντιμετωπίζει την πρόκληση να επιφέρει τη δημοκρατία σε μια χώρα η οποία εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ φτωχή και να χαρακτηρίζεται από ανισορροπίες. Μια χώρα όπου τον τελευταίο καιρό υπήρξαν πολλές δημοκρατικές ανατροπές. Ο πρόεδρος ε, έχει επανειλημμένα επαναλάβει ότι η κυβέρνησή του θα καταβάλει ιδιαίτερες ε, προσπάθειες για να ενισχύσει ε, τους ε, οικονομικά δύναμους. Αυτό εξάλλου είναι και ο άξονας της κοινωνικής του πολιτικής. Η κυβέρνησή του θα λάβει θα αναγκαστεί να λάβει σημαντικά μέτρα όχι μόνο για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση αλλά και ε, για να ε, καλύψει και τα κενά ε, της οικονομικής κρίσης. Στο Ελ Σαλβαντόρ εξακολουθεί να υπάρχει βία και εγκληματικότητα. Για να αντιμετωπιστούν λοιπόν αυτές οι προκλήσεις, η κυβέρνηση χρειάζεται εσωτερική και εξωτερική βοήθεια από πουδήποτε και αν μπορεί αυτή να προσφερθεί. Η ομάδα εργασίας σε η ΓΑΜΑ ε, ε, χαιρετίζει την ε, στήριξη του Σαλβατόρ κυρίως σε την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία βασίζεται στην ασφάλεια και στην ανθρώπινη προσπάθεια το ε, πρόγραμμα ΕΝΙΠΕ, το εθνικό πρόγραμμα, το οποίο φτάνει μέχρι το 2013. Αυτό θα διαθέσει 48,4 εκατομμύρια ευρώ για δύο τομείς, για την κοινωνική συνοχή και για την ανθρώπινη ασφάλεια. Όπως λοιπόν σας είπα ήδη, οι δύο αυτοί τομείς είναι καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση της φτώχειας στο Ελ Σαλβαντόρ. Η ομάδα εργασία συμμερίζεται την στρατηγική της Επιτροπής με την έννοια ότι οι προσπάθειες αφορούν προγράμματα όπως το Προεντούκα και το Προχάβενες. Εκεί λοιπόν πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειες, οι οποίες αφορούν όχι μόνο στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, αλλά και στις ε, βασικές αρχές που συμπεριλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα. Η δική μας η ομάδα εργασίας ε, θα ήταν ευγνώμων αν η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του πρώτου προγράμματος από το 7 μέχρι το 10 όπου γίνεται λόγος για κοινωνική συνοχή, ε, για εμπόριο. Εάν λοιπόν ε, μπορούσε να μας στελεί το συντομότερο δυνατόν αυτή η εξολόγηση. Όσον αφορά ε, τις δυνατότητες χορήγησης βοηθείας, η ομάδα εργασίας θεωρεί ότι μέχρι τώρα έγινε πολύ καλή εκμετάλλευση των, της πολύ, πολύ σωστή χρήση της βοήθειας της δημοσιονομικής. Εκτός λοιπόν από πολύ καλά ενσωματωμένες πολιτικές, ε, αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι να συμμετέχουν στις δραστηριότητε και ε, το ε, κοινοβούλιο και η κοινωνία. Θα ήμασταν λοιπόν ευγνώμονε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορούσε να μας δώσει το των δυνατόν πληροφορίες για το ποιο ακριβώς ήταν ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και του Κοινοβουλίου ε, και πώς αυτοί συνέβαλαν στην επιτυχία του εργαλείου. Η δική μας η ομάδα εργασίας ε, χαιρετίζει ε, τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου λαμβάνονται υπόψη όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς. Επίσης επιθυμούμε να προσθέσουμε ότι η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να καταλήγει ε, σε κάτι απλά τυπικό. Γι' αυτό λοιπόν ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να αυξήσει, να εντείνει τις προσπάθειες έτσι ώστε τόσο η κοινωνία των πολιτών όσο και το, το, Κοινοβούλιο να συμμετέχουν στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Συμπεράσματα. Έχουμε τρία βασικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των στρατηγικών εγγράφων. Καταρχήν, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι τα μέτρα τα οποία προτείνει η Κομισιόν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Πρόκειται λοιπόν για την επάρκεια των μέτρων ε, σε τομείς ε, μεγάλης ε, στρατηγικής σημασίας. Εκτός αυτού, Όλα αυτά ε, αντιστοιχούν σε ανάλυση από πλευράς ε, της χώρας ε, και της Κομισιόν. Δεύτερον, όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο που προέκυψε μετά τις τελευταίες εκλογές. Το πλαίσιο αυτό μπορεί να προσφέρει νέο ενθουσιασμό για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια στη χώρα. Η δική μας ομάδα εργασία αναγνωρίζει ε, πόσο δύσκολο είναι να εργάζεται κανείς σε ένα τόσο ευαίσθητο πλαίσιο, κυρίως ε, διότι εξακολουθεί να μένεται η κρίση. Ε, καλείται η Επιτροπή να προάγει κάποια πλεονεκτήματα της χώρας. Ποια είναι αυτά τα πλεονεκτήματα. Πρώτον, η ευθύνη υπευθυνότητα την οποία έδειξαν ε, ε, οι ντόπιοι στην ανάπτυξη της χώρας. Ε, στηρίχθηκε ο προϋπολογισμός και επίσης η κυβέρνηση ανέλαβε τη δέσμευση να καταπολεμήσει την φτώχεια και να την βάλει ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Κατόπιν επιθυμούμε να υπάρξει επισήμανση όσον αφορά την πολιτική συνοχή της αναπτυξιακής βοήθειας. Σε κανένα από τα έγγραφα εθνικής στρατηγικής που αναθεωρήθηκαν μέχρι τώρα, ε, πουθενά δεν γίνεται ανάλυση ανάμεσα στη βοήθεια που χορηγείται και στις υπόλοιπες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μας ε, η ομάδα γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι αδύνατον να υπάρχει απόλυτη συνοχή. Και θα θέλαμε να επενθυμίσουμε ότι ε, το άρθρο 208 της Λισαβόνας προβλέπει ότι όλα αυτά είναι υποχρέωσή μας και από τώρα ε, και στο μέλλον θα ήταν υποχρέωσή μας να στηρίξουμε την πολιτική συνοχή. Άρα αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να μην υπάρχει κανένα είδου ένσταση όσον αφορά αυτό το έγγραφο, όσον αφορά την ε, εθνική στρατηγική του Σαλβαδόρ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Οι συνάδελφοι, συμφωνείτε με αυτά που είπε ο κύριο ε, Γερέρο. Ωραία, είναι αυτή η περίπτωση. Θεωρώ ότι αυτά τα, αυτά τα συμπεράσματα, αυτές οι συστάσεις εγκρίνονται από την Επιτροπή μας και εδώ θεωρώ όταν ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία που αφορούσε την διαδικασία του δημοκρατικού ελέγχου και θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκέρενς ε, εκ μέρου της ε, ομάδας εργασίας ΔΕΛΤΑ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στις 4 Μαΐου ε, συναντηθήκαμε ώστε να μπορέσουμε να, να κάνουμε έναν απολογισμό σχέση με το ε, τι γίνεται όσον αφορά τη Χιλή, Παραγουάη, γιατί όσον αφορά την Χιλή, ο εισηγητής, ο κύριος Αλσπένσον δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα εδώ η κυρία ε, Οντή. Και μου ανέφερε το να κάνω εγώ την, την, ε, την παρουσιασή του και, και βεβαίω έχουμε 34 σημεία στα οποία καταλήξαμε και θεωρήσαμε ότι είναι το πιο σωστό, ούτω ώστε να μπορέσουμε να τα εξετάσουμε στην Επιτροπή μα. Ε, η κατάσταση είπαμε ότι είναι πάρα πολύ ε, συγκεκριμένη. Πρόκειται για μια χώρα που έχει πάρα πολύ προχωρήσει όσον αφορά την ε, οικονομία τη και δεν ξέρουμε τώρα κατά πόσον είναι το πιο σκόπιμο να συνεχιστεί η ενίσχυση. Και γενικότερα για όλε τι χώρε που έχουν προχωρήσει αντί την Χιλή. Ε, Επίση, πρέπει να σα πω ότι η Γερμανία, η Ισπανία αλλά και η Σουηδία ήσαν οι τρει ε, δανειστέ, δωρητέ προ την Χιλή, ε, οι οποίε μία μετά την άλλη αποσύρθηκαν. Επομένω, το θέμα το οποίο ε, τίθεται είναι τι θα κάνουμε μετά το 2013 γιατί βεβαίω έχει προταθεί το να συνεχίσει να τρέχει το πρόγραμμα αυτό που υφίσταται την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, αλλά μετά το 2003 θα πρέπει να δούμε, μπας και πρέπει να κάνουμε κάτι το νέο. Και αυτή η πρόταση τη συνέχιση της βοήθειας εκ μέρους της Κομισιόν ε, ενισχύεται αυτή η άποψη από το ότι όλη αυτή η ενίσχυση της Κομισιόν στα πλαίσια προγράμματος το οποίο ενισχύζουμε ανταποκρίνονται ε, στον κώδικα του ΟΣΑ όσον αφορά την αυξιακή βοήθεια. Όλα αυτά τα οποία έχει πει η Κομισιόν, όλα αυτά αφορούν την αυξιακή βοήθεια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε μήπως δεν χρειάζεται, δεν πρέπει πια να συνεχίσουμε αυτή μας την ε, πολιτική. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι όλοι να προβληματιστούν με αυτή τη συνεργασία νότου-νότου. σε σχέση με την τοποθέτηση των βορείων χωρών και μετά τις 2013 να θεωρηθεί service provider η Χιλία και να προσκληθούν και να εισφέρουν και αυτοί την εμπειρία τους ε, σε αυτή τη διαδικασία που την έχουμε ονομάσει τριγωνική συνεργασία αυτά για τη χιλή, επομένως προτείνουμε να μην συνεχιστεί η σχέση της συμφωνίας, όμως επειδή βάσει των θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε το 2013 όσον αφορά τώρα την Ουρουγουάη Εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ένας στους πέντε στη χώρα αυτή βρίσκεται κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Έχουμε αυτό το πρόγραμμα για την Ουρουάη και προβλέπει 17 εκατομμύρια ευρώ για τη σχετική περίοδο. Άρα θα πρέπει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Επίσης, θα πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για οικονομική ανάπτυξη. Οπότε ούτε εδώ υπάρχει καμία ένσταση, όσο δε αφορά την Παραγουάη, εκεί υπάρχουν κάποιοι κλάδοι προτεραιότητας που καλύπτουν το πρόγραμμά μας. Επίσης έχουμε και την παιδεία και από την άλλη μεριά έχουμε την οικονομική ολοκλήρωση. Είναι δύο τομείς προτεραιότητας και χρειάζεται επίσης να ενισχύσουμε την καταπολέμηση της φτώχειας σε σχέση με το κονδύλιο των 20 δις Αύξηση 10 δις προβλέφθηκαν επίσης, ώστε να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε αυτά τα 60 εκατομμύρια, δηλαδή τέσσερι φορές περισσότερα από όσα είχαν προβλεφθεί για την χιλή. Οπότε το ποσό αυτό υλοποιεί τα όσα έχει εξαγγείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την καταπολέμηση τη φτώχεια. Επίσης, είχαμε πει ότι θα πρέπει να εξεταστεί μια ε, οικονομική υποστήριξη όσον αφορά την ε, φορολογική μεταρρύθμιση στην ε, Ουρουγουάη. Και για να είναι βάσιμη τέτοια ενέργεια θα πρέπει κάθε χώρα να μπορέσει όχι μόνο να φροντίζει τα των εισοδημάτων, αλλά θα πρέπει να φροντίσει την διανομή και αναδιανομή του κεφαλαίου, τόσο ώστε να μπορεί να θεωρήσουμε ότι ανταποκρίνεται στι αρχέ τη κοινωνική δικαιοσύνη. Άρα να έχουμε μια τέτοια επανεξισορρόπηση που θα ακολουθήσει αυτή την ε, αναδιανομή του κρατικού κορβανά. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό για την Παραγουάη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν ε, ωφελεί συνέχεια να ενισχύει την κρατική για την ε, ανάπτυξη. Αυτό έτσι καλώς πρέπει να γίνει, αλλά θα πρέπει παράλληλα να δούμε κατά πόσον έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη σε μια χώρα με αυτά τα χρήματα. Και να μπορεί αυτή η χώρα και να δημιουργήσει περισσότερο εισόδημα, περισσότερο πλούτο, αλλά και να τον αναδιανέμει. Και βέβαια για προς αυτή την προσπάθεια θα κινούμε στα πλαίσια σχέση σε Αυτά όσον αφορά αυτές τις τρεις ε, χώρες, αυτά τα τρία προγράμματα, τα υποεξέταση. Άρα, να ληφθούν υπόψη, είπαμε, το τι θα γίνει μετά το 2013. Και η πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς την Επιτροπή μας μάλλον, είναι να εγκρίνει τα συμπεράσματα όπως σας τα εξέθεσε πρόεδρος. Σε ευχαριστούμε. Υπάρχουν παρατηρήσεις σε σχέση με την εισήγηση Γκέρενς. Ευχαριστώ πρόεδρε, ο κ. Γκερέρα. Όχι, δεν θα πω τίποτα για την εισήγηση Γκέρενς. Αλλά Ήθελα να πω κάτι για την ε, συζήτηση η οποία έγινε ε, σε σχέση με την ανάλυση της ε, έκθεσης. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σχετίζεται με την πολιτική ανάπτυξης την επαύριο, τι θα γίνει δηλαδή μετά το 2013, γιατί έχουν πάρα πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής που δεν μπορούν να θεωρηθούν χώρες αναπτυσσόμενες. Ούτε οι ίδιες δεν θέλουν να θεωρούνται τέτοιες και ονομάζονται χώρες σε φάση μεταβατική. Φερρυπίν η Βραζιλία. Είναι τελικά δωρητές οι ίδιες. Επομένως υπάρχουν πάρα πολλές χώρες Λατινική Αμερική οι οποίες ε, έχουν στο εσωτερικό τους ανισότητες και κοινωνικές και εδαφικές. Επομένως, σε σχέση με τα όσα μας είπε ο κύριος Γκέρν, σε σχέση με το τι θα κάνουμε στο μέλλον, ίσως θα πρέπει να δούμε και αυτή την πτυχή. Συνοχή εδαφική και κοινωνική. Και έτσι να πάμε στον καθορισμό της πολιτικής της ανάπτυξης για τις χώρες του μεσαίου σωδήματος, γιατί αυτές οι χώρες μπορεί να μην έχουν πρόβλημα γενικότερο κατά τις στόχες. Όμως, όμως υπάρχουν κάποια, κάποια κομμάτια της κοινωνίας, κάποιες μειονότητες, κάποιες περιοχές που αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι με τίποτα να μην ε, σταματήσουμε την πολιτική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Θεωρώ λοιπόν ε, ότι υιοθετήθηκαν τα συμπεράσματα από την Επιτροπή. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να σχολιάσει τις, τις παρατηρήσεις των ομάδων εργασίας C και D. και Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Συμφωνούμε με τα σχόλια τα οποία έγιναν από την Επιτροπή Αναπτύξεως και θα ήθελα να καθησυχάσω τα μέλη της Επιτροπής ότι τα στοιχεία που ζήτησαν, δηλαδή την αξιολόγηση του προγράμματος για το El Salvador θα διατεθούν εν ευθέτω χρόνο διότι καταρτίζονται ακόμη. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω το σχόλιο που έγινε σχετικά με την περαιτέρω σκέψη για την συνεργασία όχι μόνο με τη Λατινική Αμερική αλλά με όλες τις υποανάπτυξη χώρες σε βάση της προοπτικής του 2013. Είναι μια διαργασία που ξεκινά. Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας και ε, θα τα λάβουμε υπόψη. Πρόκειται να είναι μια μακρά συζήτηση και νομίζουμε ότι είναι κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσουμε. Γενικώ σας ευχαριστώ για τα σχόλια και για το πρόγραμμα το οποίο έχετε παρουσιάσει. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, το 7β όπου θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων για την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, της Νομικής Επιτροπής για τους νέους κανόνες επιτροπολογίας και την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ε, Νομική Επιτροπή εκπονεί μία νομοθετική έκθεση βάσει ε, του, των εξελίξεων που προβλέπονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα αντικατασταθεί λοιπόν η παλιά απόφαση σχετικά με την επιτροπολογία και αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητά μας δημοκρατικής εξετάσεως Πρέπει τώρα να καθορίσουμε ε, ποιοι θα είναι οι ε, κανόνες για ε, την δημοκρατική αυτή δυνατότητα εξετάσεως και ορισμένες προοπτικές οι οποίες θα καλυφθούν από θέματα που εξετάζει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Γι' αυτό και οι συντονιστές αποφάσισαν την περσμένη Τρίτη για την Επιτροπή ανάπτυξη να εκπονήσει μία γνωμοδότηση σχετικά με την έκθεση Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων διότι οι συντονιστές ήταν πεπισμένοι ότι η Επιτροπή μας θα μπορούσε να προωθήσει το σχέδιο γνωμοδοτήσεω τη προτού διατεθούν όλες οι μεταφράσεις. Ο, ομιλητής μας είναι ο Γκάι Μίτσελ και του δίνω το λόγο για 10 λεπτά. Έχετε το λόγο κύριε Μίτσελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με συγχωρείτε που άργησα λιγάκι ε, διότι ήμουν σε μια άλλη επιτροπή. Ε, θα ήθελα να σας πω καταρχήν ότι ο κανονισμός DCI και όλα τα άλλα εξωτερικά εργαλεία χρηματοδοτήσεως όπως και το μέσο χρηματοδοτήσεως για σταθερότητα ε, η επιστημιστική βοήθεια και όλα τα θέματα λειτουργούν επί της ιδίας λογικής. Δηλαδή δηλαδή ε, η Επιτροπή και το Συμβούλιο καθορίζουν την μακροπρόθεσμη πολιτική ε, εν αντιθέσει προς τα θεματικά έγγραφά μας και μετά υπάρχουν διατάξεις σε ενδεικτικά ε, πολιετή προγράμματα και μετά στα συγκεκριμένα προγράμματα. Όπως γνωρίζετε ελέγχουμε αυτά τα μέτρα ιδίως για να αποφύγουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραβεί τους βασικούς κανονισμούς, να υπερβεί τις δυνατότητές της και τις αρμοδιότητές της και ε, να εφαρμόσουμε και τις δυνατότητες του Κοινοβουλίου σε, αυτά, σε, αυτό το τομέα. Ε, διότι ε, πρέπει να προχωρήσουμε. Ε, οι κανόνες όσον αφορά ε, τις ε, αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου βασίζονται στην Επιτροπολογία έχουν αποφασιστεί από το Συμβούλιο χωρίς τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και η συνθήκη της Λισαβόνας έχει αλλάξει άρδιν το σύστημα της Επιτροπολογίας το οποίο τώρα καλύπτεται από δύο κατηγορίες δράσεων. Καταρχήν κατανάθεση και δεύτερον εφαρμοστικές ε, δράσεις όπου ε, η εφαρμογή γίνεται από τα κράτη-μέλη μόνο και γι' αυτό στην μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση ε, της DCI ε, η Επιτροπή είναι συσπηρωμένη και επιμένει ότι ε, θα πρέπει όλες οι κατανάθεση δράσεις να βασίζονται σε προγράμματα και τα προγράμματα δράσεως να καλύπτονται από τις διατάξεις για τις εφαρμοστικές δράσεις και όλες να θεωρούνται εφαρμοστικές ε, δράσεις και ως εκ τούτου το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, καθορίζει τις προδιαγραφές. Ε, όπως ελέγχθη η Νομική Επιτροπή εκπονεί μία νέα πρόταση για την επιτροπολογία διότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προβλέπει καμία δράση του Κοινοβουλίου δεν και θα έπαιρνε τα έγγραφα στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τη στρατηγική την εποχή που θα τα έστελνε και στις χώρες τις εμπλεκόμενες. Πράγμα το οποίο ε, δεν ε, συνάδει με ε, τη νομοθεσία. Χρειάζεται λοιπόν μία οριζόντιος ευθυγράμμιση όλων των δράσεων εκτός της ε, κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο επί της οποίας δεν έχουμε επιτύχει ακόμη. Δηλαδή όλη η επιτροπολογία για τα εξωτερικά εργαλεία χρηματοδότησης ε, θα μπορούν ε, να εξεταστούν εκ προημίου και γι' αυτό η εφαρμογή εφαρμογή η εφαρμογή των εφαρμοστικών ε, ε, ενεργειών ε, δεν πρέπει να προεξοφλήσει τα, ότι θα απεμπολίσουν τα δικαιώματά μας να εξετάζουμε τη διαδικασία να πάσα στιγμή στο μέλλον και πρόκειται για μία πρόταση με την ε, τακτική διαδικασία, δηλαδή συναπόφαση. Άρα το Κοινοβούλιο μπορεί να την τροποποιήσει εάν ε, ε, παραμείνουν στις θέσεις τους οι συνάδελφοι της Νομικής Επιτροπής για να διατηρήσει το Κοινοβούλιο το δικαίωμα δημοκρατικής εξετάσεως, πρόσβασης στις πληροφορίες και να τις ενισχύσει εφόσον τώρα υπάρχει συνθήκη της Επιπλέον θα προτείνω και τροπολογίες για να ε, ε, ε, δώσω νέες δυνατότητες και νέες εξουσίες για να μειώσουμε την την ε, ε, τις επιπτώσεις ε, των μονομερών δράσεων. Δεν ξέρω όμως η νομική επιτροπή, η επιτροπή τι θέση θα πάρει στο θέμα αυτό και γι' αυτό θα πρέπει να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μας χωρίς εμπόδια και ελπίζω ότι θα με στηρίξετε και τώρα και στο μέλλον για να ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχουν ε, οι ευρωβουλευτές εάν ε, το επιθυμούν ή ο κύριος Πένικτον, ο, κύριο, ο κύριος Ντεβά καταρχήν. Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να ακούσω πολύ προσεκτικά αυτά που είπε ο φίλος και συνάδελφος κύριος Μίτσελ και με απλά λόγια. Ερωτώ, η συνθήκη της Λισαβόνας μας ε, προσφέρει ε, περισσότερες δυνατότητες ελέγχου ή περισσότερες δυνατότητες λήψης αποφάσεων. Γιατί ε, το ένα είναι σαν να εποπτεύει κανείς τη δουλειά κάποιου άλλου και να κάνει τα σχόλιά του. Το άλλο είναι το να έχει κανείς αρμοδιότητες στο να συντάσει την νομοθεσία. Πρέπει να πω ότι αντί να μιλάμε για διαδικασίες λήψη αποφάσεων, μιλάμε περισσότερο για διαδικασίες ελέγχου, εκτός αν δεν κατάλαβα καλά. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Γκέρενς. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας πω εκ προημίου ότι συμφωνώ με τα συμπεράσματα τα οποία προτείνει ο συνάδελφος κύριος Μίτσελ. Βεβαίως θα ήθελα να ακούσω τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, επί του θέματος και νομίζω ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να μειωθεί το δικαίωμα το οποίο έχουμε εξασκήσει μέχρι στιγμής και να μην μπορούμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της mid-term review. Διότι εμείς δεν ενοχλούμε, συζητάμε ανοιχτά και ειλικρινά για τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζονται τα προγράμματα και προσπαθούμε να συμβάλλουμε στη λύση και όχι να διονγκώσουμε το πρόβλημα. Επίσης η αξιολόγηση είναι ένα μέρος του κύκλου προγραμμάτων. Εάν σε ένα σωστό πρόγραμμα, εάν δεν περιληφθεί η διάσταση της αξιολόγησης, τότε ε, στερείται από ένα βασικό εργαλείο για να μπορέσει να ε, έχει διάρκεια και σταθερότητα αναπτύξεως και από αυτού θα ήθελα να αναφέρω ορισμένε σκέψεις πολιτικές ε, τις οποίες έχω κάνει και που θα συμπληρώσουν ε, τις σκέψεις του κυρίου Μίτσελ. Θα ήθελα όμως πρώτα απ' όλα να ακούσω τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ζητώ να μου απαντήσει και σε ένα δεύτερο ερώτημα. Είναι γενική άποψη της Επιτροπής Μπαρόζο που εμποδίζει ενδεχομένως να προσεγγίσει την Επιτροπή μας. Μου φαίνεται, μου φαίνεται πιθανό. Αυτό που μου φαίνεται μάλλον απίθανο είναι να πρόκειται για ένα διάβημα της Γενικής Διευθύνσεως Αναπτύξεως και Συνεργασίας και του Επιτρόπου Πίμπαλτς. Δεν θα μπορούσε να έρθει ο κύριος Πίμπαλτς ε, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, το οποίο είναι πολύ πολιτικό. Και εφόσον στήριζε την προσπάθειά μας, νομίζω ότι καλό θα ήταν να συγκλίνουν ε, οι απόψεις μας για να μπορέσουν μπορέσουμε να εξετάσουμε δημοκρατικά ό,τι γίνεται στο θέμα των DCI. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μάρτιν Πένιγκτον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο κύριος Μίτσελ, ότι δηλαδή η Κομισιόν έχει καταθέσει δύο προτάσεις, η μία αφορά την εφαρμογή του 290 της συνθήκη της Αβώνας και η δεύτερη αφορά το 291. Αναφέρθηκε στο ότι κατά το παρελθόν οι επιτροπές επέμειναν ότι η Κομισιόν θα πρέπει να τηρήσει τους όρους του DCI και μάλιστα θέσψε και διάφορα ψηφίσματα επ' αυτού. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εμείς ε, προσπαθήσαμε όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας ε, καταθένοντας ε, προτάσεις για τα εργαλεία και της ενδιάμεσης αναθεώρησης και θεωρούμε ότι οι αλλαγές στα εργαλεία θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου. Επίσης νομίζω ότι η συζήτηση που μόλις τώρα είχαμε σε σχέση με το δημοκρατικό έλεγχο και τις συζητήσεις για τα έγγραφα της διάμεσης αναθεώρησης Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ένας ζωντανός διάλογος και επίσης ότι η Επιτροπή ενδιαφέρεται να ακούσει τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου ε, σε σχέση με τις προτάσεις για τις διάφορες χώρες. Επίσης αυτό που είναι σημαντικό είναι το Κοινοβούλιο να τα όλα αυτά υπόψη του. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρόκειται για διάλογο κοφών. Απλά ε, τώρα το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο μπορούν να συνεχιστούν οι συζητήσεις για τις προτάσεις τις οποίες έχει καταθέσει η Επιτροπή. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό ε, να μείνει αυτή η αρχή της ε, αυτόματης αναπροσαρμογής. Εμείς πιστεύουμε ότι το σύστημα της επιτροπολογίας το οποίο προσφέρει ε, πάρα πολλές προτάσεις κάθε χρόνο, το σύστημα αυτό θα πρέπει να ε, μπορεί να προχωρήσει χωρίς πρόβλημα. Και οποιαδήποτε απόκληση από αυτή την αρχή ε, θα πρέπει να είναι δύσκολη. Κατά τα άλλα, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν και άλλες συζητήσεις από αυτού. Ε, κατά την άποψή μας πρόκειται για ένα οριζόντιο θέμα που αφορά στις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της συνθήκης. Ε, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ε, δεν μπορώ να ε, τοποθετηθώ σε αυτή τη συζήτηση που μπορεί να γίνει μεταξύ κυρίου Μπέρονης και Πίπατς, αλλά εγώ θέλω, ήθελα να σας μεταφέρω τη δική μας τη γνώμη και να ακούσω ενδεχομένω και τη δική σας, αν σε αυτό το επιθυμεί η Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Merci Ευχαριστώ δεδομένου ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να καταρτήσουμε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης η προθεσμία για τις τροπολογίες θα είναι την Παρασκευή 14 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 2 Ιουνίου τώρα έχω το λόγο στον κύριο, δίνω το λόγο στον κύριο Γκάι Μίτσελ για να κλείσει ο κύριος Ντέβα Α, όχι, δεν ανεχώρησε, με συγχωρείτε, νόμιζα ότι ανεχώρησε. Θα σας έλεγα ότι ξεκινάτε ε, προς την Downing Street, αλλά σας βλέπω εδώ. Καταρχήν λοιπόν πρέπει να ρωτήσουμε αν ε, ε, η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει δυνατότητες μεγαλύτερης νομοθεσίας. Ναι, αλλά όχι για εμάς. Ήδη έχουμε μεγάλες αρμοδιότητες αλλά το θέμα είναι ε, οι ε, ενέργειες κατανάθεση όπου έχουμε ε, η δημοκρατικό δικαίωμα εξέτασης και το θέμα είναι τι γίνεται με τις υπουργικές αποφάσεις και οι οποίες ενδεχομένως δεν χρειάζεται να πληράσουν από το κοινοβούλιο οπότε για τις κατανάθεση ενέργειες σημαίνει ότι όλα θα αφαιθούν στο Συμβούλιο που θα θεωρεί ότι είναι εφαρμοστικές διατάξεις και δεν θα ενημερωνόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν ε, να θεωρήσουμε ότι η ε, κατανάθεση εργασίες είναι εφαρμοστικές, ε, ενέργειες είναι εφαρμοστικές. Δεν θέλουμε να καλύψουμε τα πάντα, αλλά θέλουμε όλα τα θέματα να έρχονται στο Κοινοβούλιο και να, θα πρέπει να έχουμε και νομικά αυτή τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα και χαιρετίζω τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να μας προσεγγίσει και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Αλλά δεν είναι ένα σημείο από το οποίο μπορούμε να κάνουμε πίσω, είναι μονόδρομος και θα πρέπει ε, για όλα αυτά τα θέματα να προχωρήσουμε. Δεν θέλουμε να ε, ε, επιβραδύνουμε καμία διαδικασία, αλλά το Κοινοβούλιο είναι Κοινοβούλιο, είμαστε νομοθέτες, πρέπει να μας λαμβάνουν υπόψη και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συζητήσει μαζί μας είναι εξαιρετικό ο Επίτροπος, μπορούμε να συζητήσουμε, να ξαναξεκινήσουμε τις συζητήσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, το ταχύτερο δυνατόν. Ωραία, ο κύριος Ντέβα έχει το λόγο. Άρα, έχω δίκιο. Εάν θεωρήσω ότι έχει ειλικρινές προθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά ότι έχει στόχο να συμμεριστεί αυτό το οποίο θέλει το Κοινοβούλιο και επομένω να υποστεί στον δημοκρατικό Λόγο του Κοινοβουλίου και να μην είναι επομένω αόρατη σε κάποιο που δεν είναι αιρετό. Επομένω να είναι πιο όρατη, να έχουμε κάτι πιο προβλημένο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επομένω να έχουν την εικόνα, να, να αποκτήσουν την εικόνα κάποιου πραγματικού ανθρώπου που ανταποκρίνεται. Επομένω, εάν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι έχει λοιπόν ειλικρινέ προθέσει ο Κομισιόν, τότε να θεωρήσω στη συνέχεια σαν συνέπεια που δεν έχει καμία ένσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το να έχουμε τέτοιου είδου κατανάθεση πράξη για την πολιτική μα. Αλλιώ, εάν έχετε κάποια ένσταση, τότε να θεωρήσω ότι δεν θέλετε να είστε ορατοί και να υποστείτε την ε, δημοκρατική ε, λογοδοσία και ευθύνη. Μπορείτε να μας πείτε ναι ή χωρίς να προσφύγουμε σε ανακοινώσεις τύπου. Κύριε Μπέρμα, έχετε το λόγο, λέει η χωρις να προσφυγουμε σε ανακοινώσει τυπου κυριε μπερμα εχετε το λογο λεει ο προεδρος ετσι για τα προηγουμένα να σας πω ότι η σοσιαλιστική ομάδα συμφωνεί με τον Γκέι Μίτσελ ότι δηλαδή ε, οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου δεν είναι δυνατόν να υπονομεύονται υπό αυτές τις νέες περιστάσεις. Στην Λισαβόνα έχει τελείως διαφορετικό στόχο, το πνεύμα της ήταν το ότι θα πρέπει να καταστεί δημοκρατική η Ευρώπη. Όμως δεν είναι δυνατόν να πίσω γυρίζουμε. Άρα αυτά τα οποία τρώμε λίγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απαράδεκτα. Απλώς δεν σας τα είπα πιο νωρί, γιατί θεώρησα ότι δεν δικαιούμαι μια που άργησε να ρωτώ συνεδρίαση. Κυρία Κέλλερ. εγώ θα ήθελα να καταβεί στα πρακτικά ότι συμφωνώ. Όπω ο προλαλή σα, όπω και άλλοι. Ανέκαθεν δίναμε την μάχη μα για τη συνθήκη τη Λισαβόνα και ακριβώ θεωρούμε ότι θα εκδημοκρατήσει την ΕΟΚ. Παρά τα όσα άλλα δεν μα αρέσει. Όμω κάνει αυτό το οποίο θέλουμε, δηλαδή να γίνει πιο δημοκρατική η Ένωση, η Ευρώπη. Άρα Θυμηθείτε πόσα πρεσβεύατε και όσο θέλετε να περάσετε στις κυβερνήσει σας ή στο λαό που υπήρχε δημοψήφισμα. Επομένω, θέλετε μέσω γίνεται περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο. Είναι το, το, το δικαίωμα του και η αρμοδία του Κοινοβουλίου να προβαίνει σε αυτόν τον έλεγχο. Πρόεδρο. Ίσως ο κύριος Πένιγκτον θα πρέπει να δευτερολογήσει, διότι δεν απαντήσατε, δεν άκουσατε απάντηση ίσως όσα ερωτηθήκατε.

Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Απαντώντας τον κύριο Ντέβα θα ήθελα να του πω ότι ξέρετε εγώ έχω περάσει ώρες ολόκληρε στην ομάδα εργασία για να εξετάσουμε αυτή τη στρατηγική. Υπάρχει ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Αυτό που χρειάζεται είναι ε, η νομική έρευνα, ε, η νομική διάσταση τη συνθήκη τη Λισαβόνα και πώ μπορεί αυτή να εφαρμοστεί στην πράξη. Το θέμα είναι ότι βλέποντας και εξτάζοντας τα ε, αναπτυξιακά προγράμματα νομίζω ότι όλοι ξέρετε έχουμε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα πάρα πολλές ώρες. Έχει λάβει χώρα διάλογος, ε, ειλικρινής διάλογος και αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα είναι η νομική εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης Λισαβόνας. Ο κύριος Μίτσελ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω το εξή ότι στη δική μου τη χώρα είχαμε ε, δύο δημοψηφίσματα για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, ένα πρόβλημα που δεν ε, τέθη είναι ότι δίνει περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εμείς έχουμε νομική άποψη. Και ευτυχώς το Κοινοβούλιο είναι και ανεξάρτητο. Γι' αυτό λοιπόν οι συζητήσει συνεχίζονται. Ευχαριστώ του συναντέλφου για την υποστήριξη και ελπίζω η Κομισιό να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εδώ και δυόμιση χρόνια έχουμε ε, κατορθώσει το DCI να το ε, εντάξουμε σε ένα και μόνο κανονισμό και τελικά καταλήξαμε σε μια πολύ καλή ρύθμιση. Η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικός για το Κοινοβούλιο, ε, κυρίως ε, σε εκείνες πράξεις όπου γίνεται εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, για την υποστήριξή σας και ελπίζω ότι τελικά θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική και λογική λύση. Στις 6 ώρα θα ψηφίσουμε, που σημαίνει ότι έχουμε ένα τέταρτο διάλειμμα. Παρακαλώ λοιπόν να επανέλθετε στις 6. Επειδή είχαμε υποσχεθεί ότι δεν θα ξεκινούσαμε πριν τις 6. Ήταν κάτι το οποίο έχουμε συμφωνήσει. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι Υπότιτλοι AUTHORWAVE

Nous allons commencer la session des votes et on va commencer par tester euh, le fonctionnement des machines. Bon. Λοιπόν, ε, θα κάνουμε την ψηφοφορία με τα μηχανήματα. Ε, πρέπει να δοκιμάσουμε τα μηχανήματα. Ας δοκιμάσουμε τώρα τα μηχανήματα. Λέμε, ξεκινάει η ψηφοφορία. Προσπαθήστε να ψηφίσετε. Ψήφισαν όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Ωραία, λειτουργεί το σύστημα. Ε, ψηφίζουμε καταρχήν την ε, γνωμοδότηση για το Αφγανιστάν. Κάποιος έχει πρόβλημα? Ίσως ψάχνετε την ε, κάρτα σας ψηφοφορίας. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για το Αφγανιστάν ε, με ανάταση χειρός, όχι με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για την τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία. Ε, ποιος είναι ε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, πρώτη συμβιβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε το 5, 6, 7, 8 και 9 ε, όλα μαζί. Μέχρι το 9. Ψηφίζουμε το 5 μέχρι το 9 όλα μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η, η ε, προφορική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. η ε, προφορική τροφολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η γνωμοδότηση Ε, θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για τροπολογία 13. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. επειδή είναι η πρώτη φορά. Πρέπει όλοι να ψηφίσουν. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία 13. Τώρα ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση στο σύνολό της. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά. Έχουμε την ε, ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε σχέση με το G20 ε, για την προφορική ερώτηση στην Επιτροπή. Τροπολογία 1. Ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ξεκινά ψηφοφορία. Κλείνει. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Χωριστά. Πρώτο μέρος. Ξεκινά ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος. Ε, ξεκινά ψηφοφορία φέρτε όλοι, κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4, ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι, λίγοι. Εγκρίνεται. Τώρα, όπως έχει τροποποιηθεί το κείμενο, ξεκινά ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. Τώρα ε, ψηφίζουμε την, ε, ε, το ψήφισμα για το, τη συνάντηση των G20 πρώτη, πρώτη τροπολογία με συγχωρείτε όχι δεν χρησιμοποιώ το σωστό έγγραφο πρέπει λοιπόν να ξαναξεκινήσουμε Τροπολογία 12. Ξεκινά η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι, λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 13. Ξεκινά. Πρώτο μέρος. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 ξεκινά. Για το πρώτο μέρος ψηφίσατε, Λίγη; εγκρίνεται. Δεύτερο, ξεκινάει η ψηφοφορία, λίγοι, εγκρίνεται. Μα συγχωρείτε, απορρίπτεται, λέει η πρόεδρος. Τροπολογία 15. Λίγη. Εγκρίνεται. Δεκαέξι. Χωριστά. Πρώτο μέρος. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ψηφίσατε όλοι, λίγοι. Απορρίπτεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί 17, 18, 19. Ξεκινά ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, λίγοι. Εγκρίνεται. Είκοσι. Ξεκινά. Κλείνει. Απορρίπτεται. 21. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται. 22. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι απορρίπτεται 23 ξεκινά ψηφίσατε όλοι λίγοι απορρίπτεται 24 ξεκινά ψηφίσατε όλοι λίγοι εγκρίνεται 25 χωριστά. Πρώτο μέρος ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος ξεκινά. ψηφίσετε όλοι. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Ξεκινά, λίγη. Εγκρίνεται. 9. Ξεκινά. Κλείνει. Εγκρίνεται. 10. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 11. Ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα ψηφίσουμε όλα μαζί. Όχι. Τότε 26. Ξεκινά. από το 26 μέχρι το 4 μπορούν να ψηφιστούν μαζί. Ξεκινά. Κλείνει εγκρίνεται. 5 ξεκινά. Λίγη. Εγκρίθηκε. 6. Τροπολογία 6. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 7. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Και ψηφίσουμε το συνολικό κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Τώρα, να ψηφίσουμε την ε, έκθεση Τάις Μπέρμαν. Μαζί, το 1, το 2 και το 3, με ηλεκτρονική ψηφορία. Ψηφίζουμε, πρώτες τρεις ε, τροπολογίες ψήφισαν όλοι, πέρας, εγκρίνεται. Τι θέλετε. Α, δεν είναι αφορά αυτό. Ωραία. Παράγραφος υπαριθμών 5. Χωστή ψηφορία το πρώτο τμήμα. Π είναι υπέρ. Κατά. Και π. Απέχουν εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Π είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Χωστή ψηφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Όλα μαζί. Όλες μας μέχρι το τέλο Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματο. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Έκθεση Κάσμαν είναι, ναι. Εδώ. Πάρα πολύ σύντομα θα λάβει τον λόγο ο Σκιώδης εισηγητής για την έκθεση Κάσουμε. Ενάμιση λεπτό. Έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα, ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πολύ σύντομα, αγαπητοί συνάδελφοι, σας επισημάνω το γεγονός ότι μέχρι τώρα αποφύγαμε ε, να αποδώσουμε σημασία στις χώρες της Κεντρικής Ασίας ε, όπου όχι μόνο υπάρχει στενότης αλλά και ορισμένες χώρες όπως το Κυργιστάν και το ε, κατά καιρούς αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές καταστροφές. Γι' αυτό θεωρώ θα ήταν χρήσιμο να διευρύνουμε την προοπτική μας σε χώρες ε, που έχουν μεγάλα προβλήματα και στην Ευρώπη, χώρες όπως αυτή του Μόλδοβα. Ε, οι χώρες αυτές ε, δεν εμπίπτουν ακριβώς στην κατηγορία των ελάχιστα αναπτυγμένων, αλλά σίγουρα μπαίνουν στην κατηγορία των αναπτυσσόμενων κρατών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι πρέπει να διευρύνουμε το βλέμμα μας και να το στρέψουμε σε χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και ανασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα να κάνουμε την ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τροπολογία 28. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτωται. 29. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτωται. 30. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, από την Επιτροπή Βιομηχανίας ψηφίζουμε πέρας και εγκρίνεται. Από την Επιτροπή. Δεύτερη τροπολογία ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Όχι μισό λεπτό. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεν κρίνεται. 31. Ψήφισμα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 33. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτωτο. Συμβαστική υπαριθμόν 7. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτωτο. 32. Ψηφίζουμε. Καταπίπτει. Α, διότι εγκρίθηκε η συμβαστική 7. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, οπότε καταπίπτει αυτή. Άρα δεν θα ψηφίσουμε. Συμφωνούμε ότι θα καταπέσει. Συμβαστική 8. τύψη ψηφορία. Ψηφίζουμε. Πρώτο τμήμα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το 34 καταπίπτει, το 35 επίσης. 36. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτονται. 37. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 38. Ψηφίζουμε. Εδώ 39 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε. τα 14. Βιομηχανίες 14. Πέρα ψηφορίας και απορρίπτονται. 40. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ένα. 42 και 43. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική. Ε, ναι. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 45. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 46. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 47. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 48. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Σπέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. 52. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 53. Ε, Ψηφίζουμε για το 53. Ο κύριος Κάσμα ζητεί το λόγο. Πρόεδρε, εάν μου επιτρέπετε, Δεν έχουμε ψηφίσει την ε, συμβαστική 5. Εκτό μικροφώνου ο Πρόεδρος. Ναι, ναι, αυτό θα σα πρότεινα. Η πρόεδρο δεν ακούσει γιατί μιλάει εκτό μικροφώνου. Επομένω, 53. Ψηφίζουμε. Euh, le vote est clos. Donc, rejeté.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 Τροπολογία 73. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην προφορική τροπολογία. Όχι, με συγχωρείτε, 74. Ξεκινά. λίγοι Απορρίπτεται. 75. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1. Μπορώ να σας εξηγήσω εδώ την ε, προφορική τροπολογία για εν ονόματι του εισηγητή. Ε, θεωρούμε ότι θα υπήρχε τρόπος να περιορίσουμε το συνολικό αυτό ταμείο και αυτό είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο έχει ισχύσει αυτή η, η, η ε, τροπολογία. Ε, ζητούμε να ψηφιστεί σε δύο τμήματα. Ξεκινά η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ξεκινά. Λίγοι. Εγκρίνεται. 76. Ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 78 λίγη απορρίπτεται 79 ξεκινά Έχετε όλοι ψηφίσει, λίγοι. Απορρίπτεται. 80 ξεκινά λίγη απορρίπτεται 81 χωριστά πρώτο μέρος ξεκινά λίγη απορρίπτεται Δεύτερο μέρος ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 82. Πάλι χωριστή ψηφοφορία σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα κλείνει. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι, λίγοι. Εγκρίνεται. Τρίτο μέρος. Ξεκινά. Λίγοι. Εγκρίνεται. Τέταρτο μέρος. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται. Ογδόντα τρία. Ξεκινά. Λίγοι. Ψηφίσατε όλοι, λίγοι. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 3. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι, λίγοι. Εγκρίνεται. 4. Λίγοι. Εγκρίνεται. Είναι τα 13. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται. 85. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Απορρίπτεται. 86. Λίγοι. Εγκρίνεται. 87 88 το 87 καταπίπτει ξεκινά λίγη απορρίπτεται 89 λίγη απορρίπτεται 90. Le vote est ouvert. Tout le monde a voté. 90. Κλείνει. Εγκρίνεται. 91. Ψήφισαν όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται. 72. Ψηφίσατε όλοι, λίγοι. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14. Ξεκινά. Εγκρίνεται. 95. 36. Λίγη. Απορρίπτεται. 97. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη. Απορρίπτεται. 98. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη. εγκρίνεται. Συμβαστική 15 ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 101. Λίγη. Εγκρίνεται. 102. Λίγη. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 5. Ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 103. Ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. 104 ψηφίσατε όλοι λίγοι εγκρίνεται 105 ξεκινά ψηφίσατε όλοι λίγοι εγκρίνεται 106 ξεκινά λίγοι εγκρίνεται είναι τα 12 Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 107. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε ε, ε την αιτιολογική έκθεση. Τέσσερα. Έχετε ψηφίσει όλοι, εγκρίνετε. 5 και 6 μαζί. Κλείνει. Απερίφθη. 7. Ψηφίσατε όλοι, λίγοι εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά ε, απερίφθη. Συμβιβαστική 1. Ξεκινά. Λίγη. εγκρίνεται 10 10 και 11 μαζί όχι 10 λίγη απορρίπτεται 11 ξεκινά λίγη εγκρίνεται Συμβιβαστική 2. Ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται. 13. Ξεκινά. Λίγοι. Εγκρίνεται. 14. Λίγοι εγκρίνεται 15 λίγη εγκρίνεται συμβαστική τρία. ξεκινά λίγη εγκρίνεται συμβιβαστική πέντε. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη. Απερίφθη. 18. Εγκρίθηκε. 19. Κλείνει. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. 21. Θέλετε την 21 και 22 μαζί. Ε, ψηφίσατε όλοι. Κλείνει απερίφθησαν. 23. Λίγη. Εγκρίνεται. 24 μέχρι 27 όχι. 24 ξεκινά. Le vote est ouvert. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Rejeté. Απερίφθη. 25. Ξεκινά. Λίγη. Απερίφθη. 26. Λίγη. Εγκρίνεται. 27. Λίγη. Απερίφθη. Περνάμε τώρα στα εκτιμώντας. Θέλετε όλα τα εκτιμώντας να τα κάνουμε μαζί. Όχι. Ένα. Ένα, το προφορική τροπολογία 6 και 2. Όχι, πρώτα το 2. Ψηφίσατε όλοι, κλείνει, εγκρίνεται. 2. Ψηφίσατε όλοι, εγκρίνεται. ανοίγει η ψηφοφορία, κλείνει. Και τώρα έχουμε την ε, ψηφοφορία της τροποποιημένου, του τροποποιημένου ψηφίσματος. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται. Πριν φύγουν όμως όλοι, μία παρατήρηση ή ερώτηση προς τις άλλες τροπολιτικές ομάδες. Την άλλη εβδομάδα ή σε δύο εβδομάδες έχουμε στην Ολομέλεια να ψηφίσουμε την έκθεσή μας αλλά δεν θεωρείται στρατηγική οπότε δεν θα υπάρξει συζήτηση ενώ δεν νομίζω ότι η εξέλιξη του main της των φύλων είναι κάτι λιγότερο πολιτικό. Αν όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνήσουν μπορούμε να ζητήσουμε από την Πρόεδρο να πάει στην Προεδρία και να ζητήσει να χαρακτηριστεί σαν στρατηγική ε, έκθεση για να μπορέσουμε να τη συζητήσουμε. Αν λοιπόν συμφωνείτε όλοι μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Έχω κι εγώ ένα μήνυμα το οποίο ίσως δεν άκουσαν ορισμένοι από εσά στην αρχή είναι ότι έχουμε προβλήματα με την αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης. Παρακαλώ λοιπόν τους συντονιστές και τα μέλη της αντιπροσωπείας της Παλαιστίνης να παραμείνουν μετά το τέλος της συνεδριάσεως. Ο κύριος Κάσμαν και ο κύριος Μπέρμαν. Ο κύριος Κάσμαν πρώτα. Δεδομένης ε, της παρεμβάσεως του συναδέλφου νομίζω ότι και η δικιά μου έκθεση θα πρέπει να θεωρηθεί στρατηγική και να μην περιοριστεί στην ψηφοφορία γιατί είναι πολύ σημαντική και ελπίζω ότι και άλλες ομάδες θα συνενέσουν. Ο γραμματέας μου λέει όμως ότι θα πρέπει να το επενθυμίσουμε αυτό και να, επιμείνουμε σε σχέση με τις πολιτικές ομάδες. Εσείς κύριε Μπέρμαν, τι λέτε. Νομίζω ότι και η πολιτική ομάδα συμφέρει όσον αφορά τον, τον ορισμό, χαρακτηρισμό αυτής της έκθεσης στρατηγικής συμφωνώ για τη δική μου και φυσικά και επομένως συμφωνώ με αυτό το οποίο ζήτησε ο κύριος Κάσμα. Εσείς κύριε Γκέρντς και εγώ νομίζω ότι η πολιτική ομάδα συμφωνεί υποστηρίζοντας τα δύο αιτήματα των προλαλισάντων. Μπέρμαν και Κάσμαν. Και εγώ συμφωνώ. Ε, εσείς κυρία Κέλλερ τι λέτε. Εσείς θα πρέπει να ζητήσετε συζήτηση. Κατάλαβε σχέση με τον χαρακτήρα. Like this.